Buonasera. Ringrazio Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Δεν βλέπω πολύ κόσμο, ίσως το πνεύμα των Χριστουγέννων ήταν πιο δυνατό από το να έρθουν οι συνάδελφοι στην αίθουσα. Σας λέγω ότι η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται απευθείας από το ίντερνετ. Πρώτα απ' όλα θα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μετά την έγκριση περνώ στην ανακοινώση του Προέδρου. Είχαμε προβλέψει την συζήτηση του Άρθρο 70 του κανονισμού με τον κύριο Γκέρα εδώ. Στις 6 Δεκεμβρίου όμως συνάντησε ε, την Επιτροπή, συζήτησε το όλο θέμα με τους προέδρους των Επιτροπών και είχε πει ότι θα προτιμούσε σήμερα να μην συμπεριληφθεί το θέμα του στην ημερήσια διάταξη. Τώρα, αν ναι. θέλει να μας μιλήσει ο κύριος Γκερέρο για τις συναντήσεις που είχε, μπορεί να το κάνει εν συντομία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από την ε, συνάντηση με τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, συνάντησα και τους σκιώδεις εισηγητές για την έκθεση αυτή και στην συνάντηση αυτή συζητήθηκαν διάφορες δυνατότητες για να μπορέσει να κάνει στο σύνολό του το Κοινοβούλιο να ακουστεί η φωνή του πέραν των αποφάσεων που λαμβάνουν οι πρόεδροι για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εντολή κάποιας επιτροπής θα πρέπει να παρουσιαστεί και να συζητηθεί στην Ολομέλεια και ενδεχομένω να εγκριθεί, να αλλάξει. Και όπως είπε ο Πρόεδρος, εκ των υστέρων πήγα και στη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών και παρουσίασα τις βασικές γενικές γραμμές της έκθεσης. Είχα παραστεί σε μία από τις προηγούμενες συνεδριάσεις τους και μετά από την παρουσίασή μου έλαβαν το λόγο διάφοροι πρόεδροι επιτροπών συμπεριλαμβανομένου και του Ραφάλ Τσαρκόφσκι, εξ ονόματος της ΑΦΚΟ, προς αντικατάσταση του Πρόεδρου μας, και θα πρέπει να επισημάνω ότι σχεδόν ομόφωνα, άντε, ας πούμε ομόφωνα μόνο, χωρίς εξαίρεση, οι πρόεδροι των επιτροπών που έλαβαν τον λόγο είπαν ότι θα ήταν δύσκολο πολλές από αυτές τις ε, εντολές να καταλήξουν στην Ολομέλεια και να ελέγχονται συνεχώς ε, οι εντολές ε, διαπραγμάτευση κάθε επιτροπής και να παρουσιάζονται αλλαγές τι μας υπέδειξαν. Στην ΑΦΚΟ, στην Επιτροπή μας, βασικά, εμείς, εγώ στην εκθεσή μου και στο σύνολο Επιτροπή μας εκ των υστέρων, να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτρέψουμε να αποφαίνεται η Ολομέλεια, αλλά με τρόπο που στην πράξη αυτό να μην αποκαλέσει μία συνήθη πρακτική, αλλά να αποτελέσει μία, ε, σε περίπτωση επίγουσης ανάγκης, διαδικασία, σε περίπτωση που κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να θεωρηθεί η εντολή που μας έχει ανατεθεί. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ζήτησαν σήμερα να καθοριστεί η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών και μετά από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές σε μία συνάντηση της Επιτροπής μας να κάνω την επίσημη παρουσίαση της κατάστασης των πραγμάτων, να έχουμε ανοιχτή συζήτηση περί του θέματος αυτού και να καθορίσουμε την ε, προθεσμία κατάστασης τροπολογιών. Δηλαδή, συνοπτικά, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η παρουσία μου, να, να πω με την παρουσία μου στην συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών και με την συζήτηση που έγινε κυρίως εκ μέρους των Προέδρων των Επιτροπών που έχουν σημαντικό, ε, σημαντική εντολή από νομοθετικής άποψης, η άποψη ήταν να είμαι προσεκτικός ώστε να μην ε, ε, καταλήγει κάθε τέτοιου είδους εντολή διαπραγμάτευσης στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ε, Nessuno vuole intervenire. Δεν θέλει το λόγο. Ο συνάδελφος Γκερέρο λοιπόν μας είπε ποια είναι η γραμμή που θα ακολουθηθεί ώστε, ώστε να μην υπάρξουν ε, συζητήσεις επί συζητήσεων για τις διάφορες δολές διαπραγμάτευση των διαφόρων επιτροπών στην Ολομέλεια. Τώρα, όσον αφορά την ε, προθεσμία κατάσταση τροπολογιών, θα την καθορίσουμε στην επόμενη μας συνάντηση, όταν θα συζητηθεί η έκθεση. Μετά από την ε, συνάντησή μας σήμερα το απόγευμα, στην ίδια αίθουσα θα έχουμε και συνάντηση με την Επιτροπή για να συζητήσουμε από κοινού με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στις ε, διαπραγματεύσεις και κάποιοι τους είναι μέλη της δικής μας Επιτροπής, ο Μπροκ, ο Γκαλτιέρη και ο Φέρχοφστατ το θέμα αυτό. Θα έρθουν λοιπόν να μας μιλήσουν για τις συζητήσεις τις οποίες έχουν από σήμερα το πρωί και συνεχίζουν. Στις 6.30 ε, λοιπόν τους περιμένουμε. Έχει ήδη προβλεφθεί στις 9 Ιανουαρίου μία έκτακτη συνάντηση για το ίδιο θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα λεπτό και έχουμε καλέσει τον πρόεδρο Μπαγόζα και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου. Με Και όταν θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν, ε, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σημειώστε όμως την ημερομηνία της 9ης Ιανουαρίου. Στις 15 Δεκεμβρίου συναντήθηκαν και οι συντονιστές και συμφώνησαν επί του άλλου θέματος. Η έκθεση Πρωτοβουλία θα έχει διαφορετικό τίτλο, εάν συμφωνήσετε. Συνταγματικά προβλήματα της διαφοροποίησης για την ε, διακυβέρνηση της Ευρώπης. Η διαφοροποίηση, differentiation, είναι ο νέος όρος. Και θα πρέπει να ορίσουμε εισηγητή. Μετά θα πρέπει να ζήσουμε την άδεια για μια άλλη έκθεση πρωτοβουλία και μετά από αυτά που ο κ. Λαμασούρ θα έχουμε άλλη έκθεση με τίτλο «Εκθέσεις των θεσμικών οργάνων με τους εκπροσώπους Συμβουλίου που ορίζουν τα κράτη-μέλη». Οι συντονιστές όρισαν ως εισηγητή για την έκθεση αυτή τον κύριο Λαμασούρ. Πρόκειται για έκθεση γνωμοδότησης και θα περιμένουμε και τη γνωμοδότηση της νομικής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Την έχει πάρει ο, η σοσιαλιστική ομάδα την έκθεση αυτή. Δεν ε, ξέρουμε το όνομα του εισηγητού. Κύριε Γκερέρο, ξέρετε ποιο όνομα του εισηγητού. Δεν το ξέρετε ακόμη. Δεν το ξέρουμε ακόμη, λέει ο κύριος ε, Γκερέρο. Σίγουρα η κυρία Ρέγνερ. Άρα, άρα, Ρέγνερ. Εντάξει, εντάξει. Κυρία Ρέγνερ, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επί του θέματος. Έχετε λάβει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 28 Σεπτεμβρίου, της 5 Οκτωβρίου, 10 και 11 Οκτωβρίου, 24 Οκτωβρίου, 17 Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2011, πάντα. Είναι στη διάθεσή σας, όπως πάντα, εάν να, κάνει μία, να κάνετε μια παρατήρηση μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης θα θεωρήσω ότι έχουμε... και περνούμε τώρα στο πιο σημαντικό μας θέμα, το 4. Προπτικέ τη νέα θεσμικέ εξελίξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λήφθηκαν, όπω ξέρετε, από το Συμβούλιο Κορυφή του Δεκεμβρίου κάποιε αποφάσει. Πρώτα απ' όλα δεν θα υπάρξει αλλαγή της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα υπάρξει αλλαγή, επαναλαμβάνω, αντιθέτως 17 χώρες της Ευρωζώνης, 7 ή 9, δεν είμαστε σίγουροι ότι πρέπει 2 ακόμη να βουλευτούν τα εθνικές τους βουλές, αλλά 17 συν 7 ή συν 9 υπέγραψαν τη συμφωνία ή θα υπογράψουν τη συμφωνία για να μπορούμε να λαμβάνουμε κοινέ αποφάσεις. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα καθορίζει κάποιους υποχρεωτικούς κανόνες σε θέματα προϋπολογισμού. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας θα προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να κάνουμε και την διασύνδεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης, διευκρινίστη ότι δεν θα πρέπει, όπως είπα, να αλλάξουν οι διατάξεις της συνθήκης, δεν αλλάζουν, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει Και όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή οι δικοί μας οι εκπρόσωποι διαπραγματεύουν με τις κυβερνήσεις. Ελέγχθη ποιοι είναι οι δικοί μας οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε όλη αυτή την διαδικασία και θα ήθελα τώρα να ακούσω τις απόψεις σας. Διότι υπάρχουν συνταγματική ε, φύσεως θέματα που είναι σημαντικά. Δεν έχει υπογράψει η Μεγάλη βρετανική. πρέπει να δούμε ποια θα είναι οι σχέσεις πλέον της Ευρωζώνης με την Ηνωμένο Βασίλειο, με τις χώρες που έχουν υπογράψει, αλλά είναι εκτός Ευρωζώνης ή με άλλες που δεν έχουν υπογράψει. Πώς θα προσπαθήσουμε, δηλαδή, αυτή τη νέα διεθνή συνθήκη κατά κάποιο τρόπο να την εναρμονίσουμε με το κοινοτικό δίκαιο. Και σε αυτή τη διαδικασία ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τρεις συνάδελφοι που συμμετέχουν έχουν συμβολικό χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο, δεδομένου ότι υπονομικής πλευρά δεν έχουν καμία ισχύ αν θέλετε και στην προηγούμενη συνάντηση στην οποία είχαμε συμμετάσχει με τον κύριο Ζέλη, είδαμε ότι τα κράτη-μέλη ή τα, οι εθνικές βουλές έχουν κάποια εξουσία την οποία εμείς δεν έχουμε. Είμαστε όμως παρόντες για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στην ε, προπαρασκευαστική φάση και όχι στη φάση της λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα σκεφτούμε, να δούμε πέραν των εξουσιών που έχουμε, για ποιους λόγους νομικής φύσεως αν θέλετε θα πρέπει κάτι να κάνουμε και να συνεργαστούμε για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Εμείς είμαστε επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή για θέματα συνταγματικών υποθέσεων. Μας ε, βοηθά βεβαίω και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, δεν είμαστε εμεί οικονομολόγοι. Δεν μπορούμε εμεί να επηρεάσουμε την οικονομική κατάσταση, αλλά οτιδήποτε άπτεται των συνταγματικών θεμάτων είναι δική μα αρμοδιότητα. Και αυτό το προβλέπει εξάλλου και ο κανονισμό μα. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο κίνηση. Θα ήθελα να πω και δίνω το λόγο στου συναδέλφου που θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριο Ταρκόφσκι. Well, just a few κάποιες παρατηρήσεις στις ε, εξ αρχής εκ προημίου, διότι θα έπρεπε πιθανότατα να <clears throat> υπάρξουν οι άλλες παρεμβάσεις, να ακούσουμε περισσότερο πώς εξελίσσεται η συζήτηση, αλλά σε σχέση με τις συζητήσεις μας εδώ, τίνουμε να συμφωνήσουμε μάλλον ότι για να διασφαλιστεί η κοινοτική διαδικασία μέθοδός μας θα πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τα συμπεφωνημένα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσω δηλαδή προσπάθειας και στο δευτερογενές επίπεδο και η δυνατότητα επίσης να γίνουν κάποια πράγματα να ενισχυθεί η συνεργασία και να έχουμε μια λιτή συνθήκη με τα πιο σημαντικά, τα οποία διαφορετικά δευτερογενώς δεν θα γινόταν να ρυθμιστούν. Οι εκπροημίου παρατηρήσεις μου είναι ότι αυτή η συνθήκη όπως έχει συνταχθεί, έχει διατύπωθεί, εμπεριέχει κάποια στοιχεία νομίζω που και διαφορετικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας. Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τον όγκο αυτών των διατάξεων της συνθήκης. Και ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες όταν γίνεται λόγος για το συντονισμό και την προώθηση του έργου των κοινοτικών ε, θεσμικών οργάνων πρέπει να είμαστε πιο εξειδικευμένοι στις διατυπώσεις μας και για τον ρόλο του τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θα βασίσουμε τη συζήτηση μα σε αυτό το σχέδιο συνθήκη, θα πρέπει σίγουρα να προβληματιστούμε για κάποια πράγματα. Αν δηλαδή κάποια πράγματα θα πρέπει να εντάσσονται σε μια διεθνή συνθήκη ή συμφωνία ή αν θα μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά υπό την κοινοτική μέθοδο και η γλώσσα να μην είναι τόσο αμφίσιμη και γενικόλογη, οι διατυπώσεις μας σε σχέση με τα κοινοτικά θέματα. Οι πιο σημαντικές συζητήσεις νομίζω θα είναι για το ποιοι θα συμμετάσχουν, ποιοι θα υπογράψουν, θα προσυπογράψουν και αν τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης, θα αποφασίσουν ενδεχόμενα να συμμετάσχουν άμεσα ή μόνο όταν θα ενταχθούν στην Ευρωζώνη υστερότερα και τα λοιπά και τα λοιπά υπάρχουν πολλά θέματα που εκκρεμούν ακόμα. Και τέλος αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθώς συζητούσαμε κατά τη διάρκεια των συντονιστών, τη συνεδρία των συντονιστών, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αναφέρθηκε από σχεδόν όλους τους συντονιστές είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλιστεί η πρόοδος του έργου της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με τις συζητήσεις για την αλλαγή της συνθήκης. Υπάρχει κάποια τάση καμιά φορά όταν έχουμε συζητήσεις σημαντικές να δημιουργούνται ομάδες εργασίας, συντονιστικές ομάδες, ομάδες για τη στρατηγική και εμείς απλώς να ζητείτε να εγκρίνουμε χωρίς να συμμετάσχουμε σε αυτές τις συζητήσεις όταν κάνουμε λόγο για συνταγματικές αλλαγές. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί με τον τίτλο, την ονομασία της Επιτροπής μας ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρέπει να εμπλακούμε σε βάθος όταν αφορά η διαδικασία τέτοιου είδους σημαντικές αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Και για να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες θα πρέπει πιθανότατα να αναμείνουμε να ακούσουμε πρώτα τις απόψεις των εκπροσώπων μας. Ίσως εκείνοι θα μπορούν να φωτίσουν περισσότερο με τις παρατηρήσεις τους τις συζητήσεις για το σχέδιο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκουερέρο έχει τον λόγο παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκφράζω τώρα εγώ προσωπικά την προσωπική μου άποψη που όμως και αυτή βασίζεται επίσης στη θέση που κατά τους τελευταίους μήνες είχε υιοθετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας αποτελώ εγώ μέλος και η αρχική, ε, το αρχικό τμήμα αυτής της γνωμοδότησης αυτής της δικής μου σοσιαλδημοκρατικής κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ότι πιθανόν δεν, ήταν, δεν θα ήταν αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η λειτουργία, η δρομολόγηση αυτής της διακυβερνητική συμφωνίας με αυτό το συνθήκη, με αυτόν τον τρόπο. Μια και οι σημερινές ενισχύει συνθήκε προσφέρουν επαρχεί μηχανισμούς για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι που θέλουμε υποτίθεται να επιτύχουμε με αυτή τη συμφωνία. Και πράγματι είναι γεγονό είναι αρκετά γνωστό ότι η αρχική θέση τη Προεδρία του Συμβουλίου περιοριζόταν σε μια διαδικασία πολύ γοργότερη, πολύ ταχύτερη και πολύ λιγότερο αμφίσιμη όσον αφορά την ε, συμβατότητα με το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πλαίσιο, όπως με την εισαγωγή κάποιων τροποποιήσεων στο πρωτόκολλο, κάποιων τροποποιήσεων στο πρωτόκολλο υπαριθμών 12 που αφορά την ρύθμιση του υπερβολικού χρέους, ε, υπερβολικού ελλείμματος και την αντίδραση εν ώψη μιας τέτοιας κατάστασης ε, υπερβολικού ελλείμματος. Τούτου λεχθέντος οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν από πλευρά τους να δρομολογήσουν αυτή την ε, συμφωνία μεταξύ τους, αυτή τη συνθήκη εντό εισαγωγικών. Γιατί είναι συμφωνία, έτσι. Δεν είναι ακριβώς τρίτη συνθήκη, είναι συμφωνία. Δεν υπάρχει πιθανότατα μεγάλη διαφορά μεταξύ του ενός ή του άλλου, αλλά πρόκειται για μια συμβολική έννοια και σημασία και πρέπει να διαφοροποιούμε. Και μια και δρομολογήθηκε αυτή η συμφωνία, νομίζω ότι το κύριο θεμελιώδες συμφέρον της πολιτικής μας ομάδας είναι να υλοποιηθούν κάποιες από τις εξής απόλυτες προϋποθέσεις ως όροι. Πρώτον, να είναι συμβατή με τις ηθίκες αυτή η συμφωνία. Και αληθεύει ότι στο αρχικό σημείο του σχεδίου που γνωρίζουμε για αυτή τη συμφωνία όχι μόνο αναφέρεται ότι πρέπει να συνάδει και να είναι συμβατή με τις συνθήκες, αλλά αναφέρεται και ο πριτανεύων ρόλος της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων ή δικαιοδοσίας με αυτή τη συμφωνία. Και όπως λέγεται, σε αρκετά σε αρκετές διατυπώσεις ε, και γλωσσικές διατυπώσεις, αλλά ουσιαστικά με το ίδιο περιεχόμενο κάθε φορά, ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες. Αυτά λοιπόν που θα αριθμιστούν θα πρέπει να μας δώσουν την ένδειξη αν πραγματικά είναι συμβατά αυτά τα οποία ρυθμίζονται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το αντίθετο, αν υπάρξουν τριβές, μήπως υπάρξουν τριβές και ε, αντιθέσεις. Πρώτο στοιχείο λοιπόν να είναι συμβατή αυτή με τις συνθήκες αυτή η συμφωνία. Δεύτερο στοιχείο, πράγματι <clears throat> νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παράγεται με την οποία το Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να διαδραματίσει το ρόλο του ως συνομοθέτης. Αντί για μια άμεση νομοθεσία ε, σε εθνικό πλαίσιο που θα άφηνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όχι μόνο εμάς αλλά και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εκτός ε, διαδικασίας και εμπλοκής. Και το τρίτο στοιχείο, αυτό συνίσταται στο στην ουσία, στο ίδιο το περιεχόμενο αυτών των ε, διατάξεων. Υπάρχουν ομάδε σε αυτό το σώμα στην Ευρωβουλή που νόμιμο είναι και αισθάνονται ικανοποιημένε για το ότι ο προσανατολισμός αυτών των αποφάσεων στοχεύει στην δημοσιονομική αυστηρότητα και πειθαρχία, στην δημοσιονομική σταθερότητα και παγίωση και στις κυρώσεις ε, οι ποινές ε, που προβλέπονται για τις χώρες που δεν τηρούν αυτές τις διατάξεις, αυτούς τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας. Η δική μου ομάδα όπως και άλλες ομάδες του σώματος, σχεδόν όλες οι ομάδες ουσιαστικά, θα επιθυμούσαμε άλλου είδους ουσία και περιεχόμενο να αναφέρεται και να καλύπτεται που να αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σε σχέση ακόμα και με μια αναφορά στο κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης, όταν κάνουμε λόγο για δημοσιονομικές περικοπές ή πιθανές περικοπές τέλος πάντων και ε, περιορισμούς όσον αφορά ε, το έλλειμμα κτλ. Κάτι σχετικό με τον κοινωνικό τομέα και τα κοινωνικά θέματα και κάποιες από τις φιλοδοξίες, φιλοδοξίες που είχε διατυπώσει το Ευρωκοινοβούλιο να κινηθούμε προς τα ευρωμόλογα ή να μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εμπλακεί και να δράσει με κύριο ρόλο, όχι μόνο σε σχέση με την καταπολέμηση του πληθωρισμού αποκλειστικά ή για τα νομισματικά θέματα μόνο και αποκλειστικά, αλλά όπως προανέφερα να προωθήσει και την ανάπτυξη και να παρέχει κίνητρα και δυνατότητες για αυτή την οικονομική ανάπτυξη ω εχέγγυα. Άλλο σημείο το οποίο θεωρώ ανησυχητικό ουσιαστικά είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα αυτά. Αρχικά, αρχικά και σύμφωνα με τον, την αυστηρή επικέντρωση τη συνταγματικά και νομικών θεμάτων, δεν υπάρχει καμία ε, ουσιαστικά ανάγκη να εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο από ό,τι φαίνεται αυτή η συμφωνία. Και έτσι λοιπόν μας έθεσαν στο περιθώριο απλά. Εμείς δεν είχαμε τίποτα να αρθρώσουμε ως λόγο, δεν είχαμε ρόλο να διαδραματίσουμε, δεν είχαμε ψήφο και φωνή να αρθρώσουμε όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Αληθεύει ότι η εκλογή των τριών εκπροσώπων του Ευρωκοινοβουλίου που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, από κοινού με τους εκπροσώπους που θα διοριστούν από τα διαφορετικά κράτη-μέλη, συν επιπλέον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, επιπρόσθετα, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, εντάσσει, εντάσσει εντός εισαγωγικών και το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά το εντάσσει πολιτικά μόνο. Διότι δεν υπάρχει περιθώριο και χώρο για την ανάπτυξη πρωταγωνιστικού ρόλου από το Ευρωκοινοβούλιο, ενεργού ρόλου. Τώρα, σε σχέση με πτυχέ του σχεδίου που αναφέρουν στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχουν δύο πτυχέ που θα ήθελα να επισημάνω. Και με αυτέ ολοκληρώνω την παρέμβασή μου. Η πρώτη από αυτέ, όσον αφορά την δημοσιονομική διαχείριση, τα οικονομικά θέματα. Αναφέρεται και λέει ότι οι επιτροπέ ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν σχέση με θέματα οικονομικά και δημοσιονομικά θα συνέρχονται λέει σε τακτά διαστήματα συχνά ώστε να συγκρίνουν και να αξιολογούν την πρόοδο αυτής της συμφωνίας και θα το κάνουν αυτό σε συνάρτηση, ακριβώς ο όρος που χρησιμοποιείται είναι in close, close association, δηλαδή σε στενή διασύνδεση, ε, σε στενή αλληλουχία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό όμως θέτει δύο διαφορετικά μεταξύ τους προβλήματα δίνεται η εντύπωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε υποδέστερο, υποδέστερο η βαθμίδα από τα εθνικά κοινοβούλια σε σχέση με πρόσκληση σε μια τέτοια συνεδρία, σύνοδο. Και δεύτερον μπορεί να τεθεί το ενδεχόμενο να μειωθεί, να συρρυκνωθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις δικαιοδοσίες και λειτουργία του, όσον αφορά τα θέματα σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση, οικονομική διαχείριση ένα τομέα δηλαδή όπου πλήρως έχει δικαιοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορεί να τις αναπτύξει. Δεύτερη πτυχή αναφέρεται στις συνόδους του ευρώ, Euro Summits, συνόδους κορυφής για το ευρώ όπου θα συμμετέχουν αρχή κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών που έχουν προσυπογράψει αυτή τη συμφωνία, συν επιπλέον του Προέδρου του Συμβουλίου, συν επιπλέον με συμμετοχή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επισημαίνεται και λέγεται ότι θα προσκαλούνται να συμμετάσχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν υπάρχει καμία αναφορά για το Ευρωκοινοβούλιο. Καμία. Και πιστεύω ότι αν σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στο σύνολο του Κοινοβουλίου αρνούνται μια δυνατότητα να διεκδικηθεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον ένα καθεστώς προσκεκλημένου παρατηρητή που θα συμμετάσχει ακόμα και χωρίς ψήφο, δικαίωμα ψήφου, σε αυτές τις συνόδους κορυφής της Ευρωζώνης. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ευχαριστώ. Um, Ο συνάδελφος Ντάφ έχει τώρα τον λόγο. Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει πέρα από ευρύτερη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων πρέπει να είναι σαφές για μας ουσιαστικά ότι για να μπορέσει να υπάρξει σύνταξη πρόταση ψηφίσματος για την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ιανουαρίου που θα εκθέτει και θα αναφέρει τις θέσεις, τοποθετήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τους τρεις αυτούς εκπροσώπους που θα το εκπροσωπούν όσον αφορά την Task Force, ε, την ομάδα κρούσης, ε, ε, η εργασία για τη σύνταξη αυτής της νέας συνθήκης, τη διατύπωση αυτής της νέας συνθήκης, τη απουσία άλλης εντολής. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει πρώτα και κύρια να αποσαφηνίσουμε ακριβώς αυτό. Ποια θα είναι η θέση ακριβώς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς θα λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόλων αυτών. Δεύτερον, η ομάδα των φιλελευθέρων, οι φιλελεύθεροι εκφράζουν τη θλίψη τους για την έκβαση των ε, γεγονότων στο ε, Ευρωπαϊκό Αυτοσυμβούλιο που η Βρετανική κυβέρνηση η ίδια την κλασική της πολιτική για τα θέματα εμπλοκής ε, όσον αφορά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθώντας πάντα να διατηρεί μια θέση ε, στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων την ανέτρεψε και λόγω του ότι τα εσωτερικά θέματα στην στο Μεγάλο Βασίλειο συχνά έχει ε, αναγκάσει τον Πρωθυπουργό ή υπουργού να υιοθετούν μια πιο θα έλεγα ε, αποστασιοποιημένη θέση. Παρ' όλα αυτά πάντα είχαμε, συμμετείχαμε και δεν πρέπει εδώ να υποβαθμίζεται η αλλαγή πορείας της ε, κυβέρνησης ε, της Μεγάλης Βρετανίας. Η επίπτωση, η φύση, η εμβέλεια όλων αυτών σε σχέση με την Βρετανική απόφαση να θέσει αρνηση κυρία βέτο στην αλλαγή συνθήκης έναντι των 27 είναι πραγματικά θα έλεγα κέρια σημασία όσον αφορά την ε, συνταγματική ισορροπία και σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ενδυνάμει πιθανούς κινδύνους που μπορούν να διαγράφονται για την ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο και πολιτικούς κινδύνους όσον αφορά την ίδια την συνεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως διαφωνώ με τους συναδέλφους που φαίνεται ίσως να υπενήσονται και να εννοούν ότι μια διακυβερνητική συνθήκη δεν είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της ε, Βρετανικής απόφασης. Είναι νομίζω η αναπόφευκτη συνέπεια της Βρετανικής απόφασης. Και τώρα η προσπάθεια να επιτύχει το εγχείρημα κάνοντας αυτά τα οποία απαιτείται να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική, δημοσιονομική πειθαρχία από πλευράς ε, των Ευρωπαίων μέσω δευτερογενούς νομοθετικού επίπεδου και δράσης Δηλαδή όμως εδώ κάποιος, κάποιο πρωτογενές επίπεδο είναι αναγκαίο νομοθετικά και η απόφαση να προχωρήσουν με την ξεχωριστή τους αυτή πορεία είναι η ορθή. Εν πάση περιπτώσει, επίσης εκφράζω την θλίψη μου, όπως και ο κύριος Γκερέρο και εγώ, για το ότι είναι μόνο απλά μια συμφωνία για δημοσιονομική πειθαρχία και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι μια συνθήκη για μια ε, δημοσιονομική ένωση, Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Οικονομική Ένωση που θα εξέφραζε την αλληλεγγύη μεταξύ χωρών και πολιτών, κρατών μελών και πολιτών που είναι αναγκαία αυτή η αλληλεγγύη για να διασωθεί η Ευρώπη από αυτή την κρίση. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η λύση μέχρι σήμερα επαρκεί και πάει αρκετά μακριά για να επανειδρύσει μια την ε, δημοκρατική εμπιστοσύνη ε, ή την εμπιστοσύνη των ε, αγορών. Είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι επαρκής ένα ε, αναγκαίο βήμα προς τα εμπρός αλλά δεν επαρκεί. Η συνθήκη πρέπει να, είναι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να περιγράφει μόνο πράγματα τα οποία θα είναι συμπληρωματικά στο ρόλο και χαρακτήρα τους, παραπληρωματικά και συμπληρωματικά στη συνθήκη της Λισαβόνας και να μην αντιβαίνουν ή να μην είναι αντιφατικά σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας και να διευκολύνει έτσι αυτή η συνθήκη την εφαρμογή και λειτουργία των μέσων και εργαλείων και διεργασιών και διαδικασιών που ουσιαστικά προβλέπονται ως μέρος, ως τμήμα της συνθήκης της Λισαβόνας που θα, πάντα θα έχει πριτανεύοντα ρόλο και θέση όσον αφορά τις διακυβερνητικές αυτές διεργασίες μιας τέτοιας συμφωνίας το διακυβερνητικό τους χαρακτήρα. Υπάρχουν όμως και κάποια θετικά καλά πράγματα φυσικά που απορρέουν από αυτήν την πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση. Ένα κύριο από αυτά τα στοιχεία είναι ότι η συνθήκη, επειδή είναι διακυβερνητικού χαρακτήρα συνθήκη, επειδή μπορεί να υπεκφύγει, να διαφύγει την αυστηρότητα των απαιτήσεων της ομοφωνίας ε, που θα ετίθετο ως προϋπόθεση μπορεί να προχωρήσει και να ισχύει με την ε, ε, υπογραφή των όσων εγκρίνουν και προχωρούν. Αυτό είναι μια συνέπεια που θα μπορούσαμε επ' αυτής να βασιστούμε και να συναγάγουμε συμπεράσματα προχωρώντας προς τα εμπρός εν χρόνο ώστε να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Αυτό δημιουργεί όμως ένα προηγούμενο. Ένα προηγούμενο. Και θα είμαστε ανόητοι αν το αγνοούσαμε αυτό. Πολύ ελαφρόμυαλοι. Βρίσκω ότι το πρώτο σχέδιο διατύπωσης ε, αυτής της πρότασης δεν είναι πάντα σύμβατο με τα εξαπλά μέτρα, την ε, εξαπλή νομοθεσία six pack που υιοθετεί εγκρίναμε και τώρα άρχισε να ισχύει. Βλέπω και βρίσκω ότι η προσέγγιση όσον αφορά τις, ε, τις λειτουργίες και δικαιοδοσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική εξέταση, κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο τότε θα μπορέσει να λειτουργήσει εξ ονόματος των προσυπογραφώντων σαν αποτέλεσμα μια συμφωνίας κυρίων. Πράγμα το οποίο πάνω απ' όλα απαιτεί όλα τα συμβαλόμενα μέρη να είναι έτοιμα και πρόθυμα να δράσουν ως κύριοι πράγματι όλα και να είναι συνενετικά και να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Για κάποια θέματα ίσως θα βρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι περιοριστική η συνθήκη αυτή και δημιουργεί περιορισμούς μέσω αυτής της διακυβερνητικής προσέγγισης. Υπάρχουν κάποια πράγματα στο σχέδιο που δεν μπορώ να τα κατανοήσω απόλυτα χωρίς να αμφισβητηθεί χωρίς να θέλω να αμφισβητηθεί το κύρος των συντακτών αυτού του σχεδίου, ο ρόλος π.χ. του δικαστηρίου είναι ενδιαφέρον. Και αυτό επειδή γίνεται η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 273 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ στο παρελθόν προηγούμενα. Και έτσι το δικαστήριο θα πρέπει να ερμηνεύσει με αυτόν τον τρόπο, να δώσει μια ερμηνεία στην εντολή, να νομολογεί, να ε, αποφαίνεται σε περιπτώσεις που θα οδηγούνται στο Ευρωδικαστήριο μέσω προσφυγής ενός κράτους μέλους εναντίον ενός άλλου. Σε σχέση με την βάση ακριβώς ε, της έννοιας που μπορεί να ε, τη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί σε σχέση με τη συνθήκη. Είναι ενδιαφέρον αυτό σε σχέση με τον ρόλο ενός, για παράδειγμα, δικαστηρίου ε, ομοσπονδιακού χαρακτήρα. Θα συμφωνούσα με τον κύριο Γκερέρο ότι το άρθρο σε σχέση με τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων πάει υπερβολικά μακριά, ξεπερνά τα εσκαμμένα και προς την λάθος κατεύθυνση και σίγουρα αντιβαίνει και συγκρούεται με το άρθρο 121 εδάφιο 5 του 121 για τον ρόλο ακριβώς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις δικαιοδοσίες του όσον αφορά την εποπτεία και την εξέταση των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων. Και τέλος Υπάρχουν και άλλα συναφή θέματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε απόψε κατά τις συζητήσεις που θα έχουμε με τους συναδέλφους μας που θα ε, συμμετάσχουν σε αυτή, έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη συνάντηση του σημερινού απογεύματος. Τώρα, δεν υπήρξε αλλαγή δυστυχώς όσον αφορά την δικαιοδοσία, την εντολή προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο, πιο ενεργό ρόλο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης ε, από πλευράς της, που θα μπορούσε να υποστηρίξει και ενδυναμώσει, να τονώσει τις προσπάθειες ε, προς μια πιο ομοσπονδιακή διακυβέρνηση μιας πραγμαυθεντικά δημοσιονομικής οικονομικής ένωσης. Η ευκαιρία αυτή είναι κάτι που χρειαζόμαστε κατεπηγόντως και θα έπρεπε να δραθούμε αυτής. Θα πρέπει σκληρά να δουλέψουμε λοιπόν για να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγι στην πρόοδο αυτών των διαπραγματεύσεων που αν όλα πάνε καλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες ε, σύντομα. Οργά. Όμως πιστεύω ότι το ψήφισμα της Ολομέλειας της περίοδου συνόδου του Ιανουαρίου είναι ένα αναγκαίο στοιχείο που πρέπει να συμμετέχει και να ολοκληρώνει αυτή την εξίσωση σε αυτόν τον προβληματισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίως ε, για αυτή την τελευταία ε, παρατήρησή σας, η οποία είναι πολύ πρακτική. Ο κύριος Γκαργκάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και ο κύριος Γκερέρο, και εγώ θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το στάδιο εκφράζουμε κάποιες πρώτες προσωπικές απόψεις, προκαταρκτικές. Εγώ προσωπικά πριν από λίγα λεπτά είδα αυτό το σχέδιο διατύπωσης. Χθες το βράδυ δεν μπόρεσα να το διαβάσω, είχα άλλες ε, υποχρεώσεις. Το φιλομέτρησα, μια ματιά έριξα και ζητώ συγγνώμη διότι δεν μπορώ να μπω σε βάθος. Χαίρομαι διότι ο Πρόεδρος έχει συγκαλέσει συνεδρίαση για τις 9 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε θα έχουμε το χρόνο να έχουμε μελετήσει εντελεχώς το έγγραφο αυτό και θα έχουμε και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων νομίζω. Σήμερα το πρωί έμαθα για την βραδινή μας συνεδρίαση. Ε, εγώ πρέπει να γυρίσω στη Ρώμη, επομένως δεν θα μπορέσω να παραστώ ούτε σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια πολιτικά. για όλες αυτές τις θεσμικές εξελίξεις. Εμείς θα θέλαμε περισσότερη Ευρώπη βεβαίως και αυτό ανέκαθεν το υπερασπιζόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε ποιος είναι ο ρόλος που έχουμε διαδραματίσει στο παρελθόν και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτή τη διαδικασία, να την πυροδοτήσουμε, να περάσουμε από τη διακυβερνητική ε, πρακτική στην κοινοτική ε, πρακτική σε μεγαλύτερο και περισσότερο βαθμό. Και ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν θα μας χρησιμεύσει σε αυτό το εγχείρημα. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει και ο καλογερμανικός άξονας τον οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Και μάλιστα ε, θα έλεγα ότι ίσως έτσι δυσκολεύει ε, ακόμα περισσότερο η προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Ίσως φαίνεται ότι εδώ δεν εκφράζω το σεβασμό που θα έπρεπε. Ωστόσο, αυτό το κείμενο είναι ε, σίγουρα διακυβερνητικό και έτσι αλλάζει ε, το σημείο ισορροπίας στο οποίο είχαμε φτάσει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίως απουσιάζει, βεβαίως έχει υπάρξει μια διάσπαση τρόπον τεινά δεν βοήθησε το Ηνωμένο Βασίλειο από τη στιγμή που δεν θέλησε να προσχωρήσει σε αυτό το κείμενο, αλλά και από τη Γαλλία. Ε, βλέπουμε ότι είχε η Γαλλία βούληση να αποκλείσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, είναι μια διαθεσμική συμφωνία η οποία θα ε, θέσει σε δύσκολη θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι σίγουρο. Και το λέω διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαφαίνεται να έχει ουσιαστικό θεμελιώδη ρόλο από πολιτική σκοπιά. Ε, καλείται να συμμετάσχει ως εκφραστής ιδεών, αν θέλετε, αλλά όχι ε, να έχει συγκεκριμένο πολιτικό ρόλο. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τους εαυτούς μας. Τέτοιου είδους συμφωνίες αναπόφευκτα οδηγούν την επικράτηση της γαλλογερμανικής ε, συμμαχίας. Υπ' αυτή την έννοια βεβαίως χρειαζόμαστε ε, την Γερμανία, η βοήθεια της είναι πάντοτε απαραίτητη. Από την άλλη πλευρά, επίσης χρειαζόμαστε και άλλες ε, εξασφαλίσεις. Είναι ανάγκη, για παράδειγμα, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή και των αγορών στη Γαλλία, στη Γερμανία ή αλλού. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα. Και για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφεραν οι συνάδελφοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν ε, διαβάσει το σχέδιο διατύπωσης πολύ πιο προσεκτικά από ό,τι μπόρεσα εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ διαφαίνεται μια κατάφορη αντίθεση με το περιεχόμενο της συνθήκης της Λισαβόνας. Πώς μπορούμε άλλωστε ε, να καταφέρουμε ο κοινοτικός χαρακτήρας να συνεπάρχει με συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών στις οποίες μπορούν να προσχωρήσουν και άλλα κράτη-μέλη, όπως γίνεται για παράδειγμα με τη ζώνη του ευρώ. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν τη συνθήκη, ακολουθούν αυτό το μονοπάτι ε, το οποίο με πάση ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν νομίζω ότι θα μας οδηγήσει προς το σκοπό που επιδιώκουμε όλοι. Εμείς επιθυμούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα βγει τίποτα καλό από όλη αυτή την ιστορία, ούτε καν θα υπάρξουν θετικές οικονομικές εξελίξεις. Ε, κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία γιατί η προηγούμενη συνθήκη δεν ήταν ικανοποιητική. Ωστόσο, ήδη είχαμε ενδείξεις για ε, την, το απαιτούμενο δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι χώρες μέλη δεν κατάφεραν βέβαια να ε, εκπληρώσουν τις ε, προϋποθέσεις σε θέματα δημοσιονομικής πειθαρχία. Όμως τώρα φαίνεται ότι κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Ίσως καν να μην είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα γιατί δεν έχουμε την απαραίτητη θεσμική και πολιτική στήριξη η οποία άλλωστε θα εγγυηθεί ε, το νόμισμα αυτό, το κοινό μας νόμισμα. Είδαμε την αποτυχία που σημειώθηκε επί Προεδρίας πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ε, έγινε προσπάθεια τα νομισματικά προβλήματα να τεθούν πριν από τα θεσμικά προβλήματα. Ε, προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε σύνταγμα τότε και είδαμε ότι ε, επικρατούσε η προτεραιότητα η οικονομική η οποία υπονόμευε αν θέλετε τα, τις επιδιώξεις της συνταγματικές. Ε, ε, υπονόμευε το, τις κοινωτικές πτυχές της όλης υπόθεσης. Από εκεί και πέρα, ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων με έκπληξη ε, έμαθα ε, την ύπαρξη μιας έρευνας, μιας μελέτης ως προς ε, τον ρόλο των δικαστικών αρχών, των δικαστών και τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Το 12% των δικαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αγνοούν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το κοινοτικό δίκαιο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν απαντούν κάτι τέτοιο σε μια έρευνα, σημαίνει ότι πραγματικά δεν το κατέχουν το κοινοτικό δίκαιο, δεν θα απαντούσαν αρνητικά. Δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν επικρατεί το, υπερισχύει το κοινοτικό δίκαιο ή το εθνικό δίκαιο ε, και σε ποιες περιπτώσεις ε, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όταν έγιναν οι διαπραγματεύσεις με τη συντακτική συνέλευση, είχαμε ε, μία μακροχρόνια διαδικασία, πολλή δουλειά. Ε, νομίζω ότι σημειώθηκε η επιτυχία, αρκετά μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια ξέσπασε η οικονομική κρίση και έχουμε φτάσει στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι ε, γίνονται βήματα προς τα πίσω, οπισθοχωρούμε με αυτή τη συμφωνία απομακρυνόμαστε από μια πραγματικά κοινοτική Ευρώπη. Νομίζω ότι η συμφωνία αυτή είναι ένα βήμα αρνητικό προς τα πίσω και όχι κάτι το θετικό προς τα εμπρός. Να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Εγώ προσωπικώς ε, θα τα σκεφτώ επισταμένως κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπρόντς. Στην πρώτη παραγραφό αναφέρεται ότι τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή 17 χώρες μέλη του ευρώ συν ε, ενδυνάμει 7 ή 9, έχουν την υποχρέωση ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, θεωρούν ότι η οικονομική πολιτική τους είναι ε, κοινό θέμα, θέμα κοινή ανησυχίας. Από τη στιγμή που είναι συμβαλόμενα μέρη λοιπόν, θα έλεγα ότι μας εκπλήσει το άρθρο 1 21 και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν ε, το ξέρω απ' έξω. Είδα το άρθρο λοιπόν 121 της συνθήκης και βλέπω ότι εκεί όντως υπάρχει υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να θεωρούν την οικονομική τους πολιτική ως κοινοτικό ζήτημα, ζήτημα που είναι, έχει κοινοτικό χαρακτήρα και θα πρέπει να αποσκοπούν στην ευρύτερη οικονομική εναρμόνιση και όχι μόνο στην εναρμόνιση των προπολογισμών. Δηλαδή λέει κάτι το σχέδιο αυτό διατύπωσης που ήδη υπάρχει. Στη δεύτερη του παράγραφο λέει ότι ο στόχος των κρατών μελών και των χωρών των, ε, του ευρώ είναι να ενσωματώσουν τη συμφωνία αυτή στις συνθήκες που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τον 26 αλλά όχι ακόμα τον 27. Και μέχρι ότου ενσωματωθεί η συμφωνία συμφωνία αυτή ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία παραμένει, ε, ως, παραμένει με το χαρακτήρα του ιδιωτικού συμφωνητικού και όχι μέρος του κοινοτικού δικαίου. Οι αντιρρήσεις του κυρίου Κάμερον ήταν αρκετά ε, ρεαλιστικές και όχι μόνο επί της αρχής. Στη δέκατη παραγραφό λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την αναθεώρηση όλων αυτών των διατάξεων Βάσει των άρθρων 126 και 121 της συνθήκης ε, δεν έδρασε μέσα στο πεδίο των ερμοδιοτήτων της. Έχει την εξουσία και την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει την εφαρμογή μια συνθήκη η οποία δεν είναι συνθήκη αλλά είναι μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ 17 ή 23 χωρών μελών. Το άρθρο 121 και το 126 ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, ενώ το 136 εφαρμόζεται και ισχύει μόνο στις χώρες μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Στην 10η παράγραφο λέει ότι η συμφωνία θα, είναι σε, ε, θα συμμορφούνται με το 4,1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή καλύπτονται ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και όχι όλων. Και τέλος, στην παράγραφο 24 λέγεται ότι τα συμβαλόμενα μέρη, ε, αν ένα συμβαλόμενο μέρος θεωρεί ότι κάποιο άλλο συμβαλόμενο μέρος δεν έχει ε, εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα του 3,6 της συμφωνίας, μπορεί να φέρει το ζήτημα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη δικαιοδοσία να εκφέρει απόφαση και να επιβάλλει την εφαρμογή και την τήρηση ιδιωτικών συμφωνιών μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και όχι όλων. Ε, φαίνεται ότι ε, ε, ότι πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τη συγκατάθεση όσων τον παραβαίνουν τελικά. Αυτό είναι το σχολείο μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, εκτός μικροφώνου. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Λαμασού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις μου, οι οποίες είναι απολύτως προσωπικές. Λυπούμε διότι ε, ε, διάφοροι συνάδελφοι αλλά και οι συγητές δεν μπορούν να είναι παρόντες γιατί πρέπει να, να παραστούν σε άλλες συνεδριάσεις. Προσωπικά χαίρομαι με την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε ε, στη Σύνοδο Κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου. Ωστόσο, με ανησυχεί ιδιαιτέρως η νομική ερμηνεία που προτείνεται σε αυτό το στάδιο. Ξέρετε, στη, στον ταοισμό, στην κινέζικη φιλοσοφία αυτή, Υπάρχει μία συνθήκη φιλοσοφικού χαρακτήρα, όχι διπλωματικής υφής, η οποία αποκαλείται <laughs> μικρή συνθήκη του απόλυτου κενού. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτε το νομικό στο κείμενο αυτό. Κατά την άποψή μου, τα συμβαλόμενα μέρη ε, εκφράζουν υποσχέσεις, δεσμεύονται για την ανάλυση της δράσης, δεν δρούν, δεσμεύονται ότι θα δράσουν. Είτε στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας, προσφεύγοντας ε, στο εργαλείο της ενισχυμένης συνεργασίας. Χρειαζόμαστε όμως μια καινούργια, μια καινούργια συνθήκη για να πούμε ότι θα αξιοποιήσουμε μια διάταξη που ήδη έχει ενσωματωθεί στην υφιστάμενη συνθήκη. Ή τα συμβαλόμενα μέρη δεσμεύονται να εισαγάγουν νέες διατάξεις στα εθνικά του συντάγματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι η απόφαση αληθινά δεν λαμβάνεται σε αυτές τις συνθήκες, θα ληφθεί τη στιγμή της τροποποίησης των εκάστοτε εθνικών συνταγμάτων. Δηλαδή είναι μια δέσμευση ανάληψης υπόσχεσης αυτή η συμφωνία, η οποία μάλιστα δεν περιλαμβάνει καμία κύρωση. Εάν μια χώρα υπογράψει αυτή τη συνθήκη, την επικυρώσει και δεν τροποποιήσει το εθνικό του σύνταγμα στη συνέχεια, δεν έχει καμία κύρωση. Αυτό δεν είναι νομικό. συντάξαμε και θέλουμε να υπογραφεί υπό τη μορφή της συνθήκης ένα πράγμα το οποίο είναι μια υπόσχεση χωρίς κυρώσεις. Γίνεται λόγος για τη χορήγηση στα κράτη-μέλη της δυνατότητας να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Το άρθρο 273 της συνθήκης ήδη το προβλέπει. Είναι ήδη εφικτό αυτό. Αλλά ούτε εδώ θα έχουμε κυρώσεις. Εάν ένα κράτος μέλος κατατύχει να πω τη Γερμανία αποφασίσει να ε, εγκαλέσει ένα άλλο κράτος μέλος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γιατί το δεύτερο κράτος μέλος δεν ε, τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και ε, υποτίθεται ότι θα έχει εντάξει στο εθνικό του σύνταγμα. Ποια είναι η εξουσία που θα έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα μπορέσει να ε, κηρύξει ε, ανίσχυρο έναν εθνικό προπολογισμό, για παράδειγμα. Είναι περίεργο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν θα είναι σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ε, προσπαθούμε να συντάξουμε μια συνθήκη, γίνεται προσπάθεια κατάληξη σε μια συνθήκη χωρίς συγκεκριμένες κυρώσεις. Γίνεται λόγος επίσης για κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια συνθήκη πάντοτε λέει ότι ένα κοινοβούλιο έχει αρμοδιότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει ποια είναι η αρμόδια από τις κοινοβουλευτικές του επιτροπές. Καλούμε δηλαδή τις κοινοβουλευτικές, καλούν αυτοί τις κοινοβουλευτικές επιτροπές να ε, συνεργαστούν. Αυτή δεν είναι διατύπωση διεθνούς συνθήκης. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντήσει ότι δεν έχει καμία όρεξη να δουλέψει με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, δεν θα δουλέψει και δεν θα υπάρχει καμία κύρωση ε, γι' αυτό. Ε, ένα άλλο κεφάλαιο ε, αναφέρεται στη σύνοδο του ευρώ. Όλα αυτά ήδη υπάρχουν. Αν θέλουν να τα βάλουν συνθήκη, καλώς, αλλά εν πάση πτώση είναι άχρηστο. Το πιο καινοτόμο είναι αυτό που ήδη ανέφερε κάποιος άλλος συνάδελφος η δυνατότητα δηλαδή να τεθεί σε ισχύ το κείμενο αυτό τη στιγμή που θα έχει κυρωθεί από 50 συν 1 της 50 ε, 1 ε, ε, των χωρών του ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματική καινοτομία. Δηλαδή, υποτίθεται ότι εισαγάγεται ένα πνεύμα, μια νοτροτή η οποία θα επεκταθεί και σε αυτή αυτή την κοινοτική συνθήκη. Έχω την πεποίθηση ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η τελευταία συνθήκη που θα έχουμε κυρώσει ομοφόνος. Δεν θα υπάρξει στο μέλλον άλλη κοινοτική συνθήκη η οποία να κυρωθεί από ομοφόνος από το σύνολο των χωρών μελών. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτομία αυτή. Αλλά υποτίθεται ότι δεν θα εφαρμοστεί παρά μόνο σε αυτήν εδώ τη συνθήκη ή συμφωνία. Προσθέτω λοιπόν το εξή. Τι θα συνέβαινε εάν, για παράδειγμα, εννέα χώρε τη ζώνη του ευρώ, έχοντα επικυρώσει αυτή τη συμφωνία ή τη συνθήκη, ανακαλύψουν ότι ε, δύο, τρεις ή τέσσερις από αυτές τις εννιά και μάλιστα μεγάλες και σημαντικές χώρες τελικά δεν κατάφεραν να περάσουν τις απαραίτητες συνταγματικές τροποποιήσεις. Δηλαδή επικύρωσαν τη συνθήκη αλλά δεν μπόρεσαν να την εφαρμόσουν. Τι θα κάνουν οι υπόλοιπε. Επομένως, ε, αυτό το κείμενο ε, με προβληματίζει ιδιαιτέρως, δεν βλέπω σε τι συμβάλλει η συμφωνία που δίδεται στην πολιτική συμφωνία της 9ης Δεκεμβρίου έχει πολύ μεγάλη απόσταση από την ε, νομική τελικά σημασία που μπορεί να έχει το ίδιο κείμενο. Εν πάση περιπτώσει, ε, θα πρέπει ε, να γίνει δημόσια διαβούλευση σε κάποιο κοινοβούλιο ε, για όλα αυτά τα θέματα. Αξίζουν τα θέματα αυτά τη δημόσια διαβούλευση. Είτε πρόκειται για μια διακυβερνητική συνθήκη ή συμφωνία, είτε ε, δεν θα χρειαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, την επικυρώσει, δεν θα μπορέσει, παρόλο που κάποιοι συνάδελφοι κοινοβουλευτικοί βεβαίω θα έχουν ε, προσκληθεί στα συντακτικά όργανα, στα νομοπαρασκευαστικά όργανα αυτής της συμφωνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αξίζει να συζητηθεί δημοσίως το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενδεχομένως ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια και αλλού, σε άλλα τέτοιου είδους φόρουμ. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αρκεστούμε σε μια ομάδα εργασίας η οποία θα συντάξει αυτό το κείμενο χωρίς δημόσια διαβούλευση. Και τελευταία παρατήρηση από πλευράς μου και θέτω ένα άλλο ερώτημα γιατί το κείμενο αυτό ε, γεννά πάρα πολλά ερωτήματα. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν τι κάνουμε με αυτή την πολιτική πρωτοβουλία. Η διάσκεψη των Προέδρων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να αναλάβει αυτή την πολιτική πρωτοβουλία. Αν κατάλαβα καλά, αποφάσισαν το ίδιο το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο να αναλάβει την πρωτοβουλία ε, βάσει ε, των προβλεπωμένων στη συνθήκη της Λισαβόνας ώστε να ξεκινήσει η ε, εκπόνηση μιας νέας ευρωπαϊκής συνθήκης. Μιλούμε για το ίδιο πράγμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να τη συμπληρώσει αυτή τη συμφωνία, να τη βελτιώσει. Πρόκειται για μια εντελώς καινούρια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων θα πρέπει να εκφέρει μια γνώμη ε, για αυτό το θέμα για να μην έχουμε ε, ε, εγχειρήματα και δράσεις που αντιβαίνουν μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, όπως πάντα, για τις πάρα πολύ εύστοχες παρατηρήσεις σας, κύριε Λάμα Και γίνονται πάντα την κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να πείσουμε ότι δεν υπήρξε αλλαγή στη συνθήκη. Διότι πριν από 10 μέρες αποφασίστηκε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στη συνθήκη. Και υπάρχουν ακόμη στοιχεία σε αυτή τη συνθήκη που υποβίενται στην ομοφωνία. Δεν είχαμε ομοφωνία την προηγούμενη πριν από 10 μέρες και αυτό θα πρέπει να το τηρήσουμε και να μην προσπαθούμε να το παρακάμψουμε. Θα υπάρξει μία διακυβερνητική συνάντηση. Πολλές χώρες θα συζητήσουν το μέλλον του νομισματό, το δικό του, όχι το δικό μας. Τι σημαίνει διακυβερνητικό. Αυτό που σημαίνει και ίσω καταλήξει σε ένα συνδυασμό χωρών που θα επανέλθουν και θα ψηφίσουν ο μπλοκ. Διότι όντω θα αποτελέσουν μία χώρα στο τέλος, διότι ο μόνος τρόπος να έχει μέλλον το ευρώ είναι να ψηφίζεται από μία χώρα. Θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις αντιδράσεις. Αυτό δεν είναι μέρος της διαδικασίας λειψοφάσεων των κυβερνήσεων. Εμείς είμαστε ευρωβουλευτές, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε αυτή την κυβερνητική συζήτηση αυτοί οι οποίοι θα λάβουν, ε, θα πάρουν τις αποφάσεις είναι εθνικοί βουλευτές και οι κυβερνήσεις τους. Εμείς δεν θα είμαστε, ακόμη για να το προσπαθούσαμε δεν θα είμαστε παρά συζήτηση. Με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του δικαστηρίου που είναι θεματοφύλακας από ό,τι φαίνεται. Και δεν θα πρέπει να ε, αργεστεί στο κάποια στιγμή να εγκρίνει και να είναι θεματοφύλακα συνθήκων που κάποιες άλλες ομάδες έχουν εγκρίνει. Τώρα, ποιες είναι οι διαταξίνθηκες που δίδουν την εξουσία ε, στην ε, συνθήκη να χρησιμοποιείται από κάποιους εκτός των τριών θεσμικών οργάνων. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Θα δοθούν ε, γιατί δεν θα δοθούν σε μας τέτοιου είδους εξουσίες, γιατί όχι. Δίπως δεν θα πρέπει με αυτή την αιτιολογία ε, εμείς να αρνηθούμε κάτι τέτοιο να το καταστήσουμε νόμιμο. Δεν είμαι σίγουρη ότι δίκαια από τι χώρε να αποφασίσει για την νομιμότητα αυτό το οποίο αποφασίστηκε τώρα. Έγινε μια κάποια ε, αξιολόγηση για το ετήσιο κόστο για τον φορολογούμενο. Αν υπάρξει ε, διαφωνία, εφόσον διαφωνία. Και αν όχι, και ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγε ώρε αυτό θα χρειαστεί να το ξαναπώ σε μια άλλη επιτροπή η οποία θα συναντηθεί διότι έτσι εξελίσσονται τα πράγματα από ό,τι βλέπουμε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρέν, ο κύριος Ράντζελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζοντας, θα πω το εξής. Δεν μπορώ να συμμετάσχω στην κοινή συνεδρίαση αργότερα, διότι έχουμε εθνικό συνέδριο στο κόμμα μου και έχω κληθεί να ομιλήσω για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη και έχουμε και εκλογέ για τον πρόεδρο του κόμματος, άρα δεν μπορώ να είμαι παρόν μετά τις 5-5.30. Αλλά δεδομένου ότι δεν μπορώ να συμμετάσχω στην συνεδρίαση με την Οικονομική Επιτροπή, θα πω ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έβαλαν τα μέλη της, της Επιτροπής ΕΚΟΝ διαφορετική από αυτή που έβαλαν εμάς. Δεν ξέρω αν είναι θέμα πρωτοκόλλου αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό να γίνουν έτσι τα πράγματα. Θα έπρεπε να διανεμηθούν οι θέσεις 50-50. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγιναν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό έχει πολιτική και θεσμική σημασία. Διότι έτσι η, τα θεσμικά θέματα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τα οικονομικά. Ίσως αυτό εξηγεί γιατί έχουμε και συνθήκες που δεν είναι πάρα πολύ σωστά και εκλεπτισμένα νομικά κείμενα, διότι κάνουν συνθήκες οι οικονομολόγοι. Δεν έχουμε νομικά κείμενα με νομικό περιεχόμενο, αλλά με οικονομικό. Μπας περιπτώσει, εγώ σας λέω θα είμαι απόνα τη συνεδρίαση, αλλά νομίζω είναι θέμα αξιοπρεπίας της ΑΦΚΟ. Η ΑΦΚΟ και η ΕΚΟΝ θα πρέπει από τις του Κοινοβουλίου να την χάνουν της ίδιας μεταχείρισης. Δεν πρέπει πρώτα να βάζουμε τους συναδέλφους της ΕΚΟΝ και μετά εμάς της ΑΦΚΟ. Μετά. από αυτές τις συμβολικές παρατηρήσεις πρέπει να προσθέσω και να πω ότι για αυτή τη συμφωνία και τις ανησυχίες που δημιουργούνται πρέπει να πω ότι είναι μια ήπια νομοθεσία από πλευρά συμφωνίας και όχι αυστηρά νομοθετική. Δεν μπορώ να δω πώς θα επιβληθούν οι ρυθμίσεις και οι κανόνες αυτοί. Τουλάχιστον έχουν διατυπωθεί. Είναι μια πρόταση όλα αυτά, το γνωρίζω. Αυτό μου υπενθυμίζει κάτι. Μου υπενθυμίζει ένα είδος θεσμό εμπορικού νομοθετικού πλαισίου που σε σχέση με συμφωνίες είναι μια άτυπη συμφωνία μεταξύ κάποιων μεριδιούχων, μερισματούχων για να επηρεάσουν να μπορέσει να ασκηθεί η επιρροή τους στην διακυβέρνηση μιας εταιρείας, στη διαχείριση των συμφερόντων μιας εταιρείας. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό απόλυτα και είναι θα έλεγα και μεροληπτικό ή εν, εν μέρη τέλος πάντων. Αυτή είναι η δική μου ανάλυση. Αλλά μετά από τις επεξηγήσεις που θα ακούσουμε απόψε, πιθανότατα οι συνάδελφοι έχουν καταφέρει από δική τους πλευράς να κατανοήσουν καλύτερα το τι στοχεύει να γίνει με αυτά τα έγγραφα, με αυτές τις διατυπώσεις. Και έτσι αν συμβαίνει αυτό θα είμαστε σε καλύτερη θέση να σχολιάσουμε και να κάνουμε την προσπάθεια να προτείνουμε κάποιες βελτιώσεις αν γίνεται. Έχω δύο κυριότερες ανησυχίες πρέπει να πω. Το πρώτο κυριότερο μέλημά μου είναι ότι το εύρος και η φύση των κυρώσεων. Ακούσαμε πολλά για κυρώσεις <clears throat> επί μεγάλο χρονικό διάστημα, επί μήνες ολόκληρους. Τώρα, διαβάζοντας όλα αυτά δεν έχουμε κάποια άποψη Ποιε ποιες ακριβώς ε, κυρώσεις και ποινές προβλέπονται και με ποιο τρόπο θα επιβληθούν σε σχέση με την κανονική τακτική διαδικασία που θα επέτρεπε κάτι. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι το καινούριο σε σχέση με τις κυρώσεις ή μήπως υπάρχει κάποιο νέο είδος κυρώσεων που θα επιβάλλονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να διευκρινιστεί και να το θυμόμαστε αυτό ως στοιχείο. Διότι πρέπει να πω ότι ακόμα και αν συμφωνώ με αυτό το βήμα 17 κράτη της Ευρωζώνης και συνολικά 26 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν διότι όπως πολύ καλά επεξήγησε ο Έντριου Ντάφ ήταν η μόνη δυνατότητα, η μόνη οδός ως διέξοδος για να σημειωθεί πρόοδος, να προχωρήσουν 26. Εντάξει, έστω. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με κάτι το οποίο είχε πρόταθει πριν από κάποιους μήνες και που <clears throat> θα απαγόρευε την ψήφο κάποιων χωρών που θα βρισκόντουσαν σε διαδικασία παράβασης ή παραβίασης. Αυτό αντιβαίνει απόλυτα οποιαδήποτε νομική διάταξη πραγμάτων, οποιαδήποτε νομική προσέγγιση, ακόμα και σε ομοσπονδα κράτη, ομοσπονδιακά κράτη. Λοιπόν ανησυχώ πρέπει να πω κάπως για αυτά. Αν κάποιος θα μας έλεγε ότι οι κυρώσεις είναι ακριβώς αυτές που προβλέπονται ήδη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αν είναι όμως καινούργιες κυρώσεις, πρέπει να γνωρίζουμε ποιες θα είναι αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε εκ προημίου. Επίσης ανησυχώ κάπως πρέπει να πω. Ακόμα και αν δεν συμμερίζομαι την ε, άποψη, την προσέγγιση κάποιων ευρωσκεπτικιστών συναδέφων που παρενέβησαν ήδη. Πραγματικά όμως ανησυχώ όσον αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του ΔΕΚ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ΔΕΚ να μπορέσει πιο ενεργά, με ενεργότερο τρόπο, χαρακτηριστικό της ιδιότητας ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ομοσπονδιακής δομής κράτους να εμπλακεί και να προσπαθήσει να προχωρήσει με τις δικαιοδοσίες του. Όμως δύο πράγματα εδώ πιστεύω είναι επικίνδυνα ως προοπτική. Ένα, ότι φυσικά το 10 θα πρέπει να σέβεται τις συνθήκες. Είναι κάτι το αυτονόητο, είναι σαφές αυτό. Διαφορετικά θα χάσει το ηθικό κύρος, τουλάχιστον το ηθικό, όχι ε, νομικό, αλλά ηθικό σίγουρα, όχι μόνο νομικό, αλλά και ηθικό. Και δεύτερον, ανησυχώ κάπως πάλι και ανησυχώ ιδιαίτερα με την ανάμιξη του δικαστικού σκέλους όσον αφορά το πολιτικό γίγνεσθε και την πολιτική δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων. Η ανεξαρτησία των δικαστών και του δικαστικού κλάδου είναι τόσο σημαντική υπόθεση που κανονικά ένα δικαστήριο δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνει και να αναμειγνύεται σε πολιτικά θέματα, πολιτικά ζητήματα. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος μια ναι, και με αυτό το κείμενο δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για οτιδήποτε, εντάξει, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος κιόλα. αν εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, δεν έχουμε ένα είδους πολιτικής ανάμειξης ή συμφυρμού πολιτικού, θα έλεγα σε σχέση με ένα συνταγματικό, συνταγματικό δικαστήριο και αυτό όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες τις δικαστικές του 10 εδώ δύο λοιπόν πτυχές ως παρατηρήσεις από πλευράς μου που θέλω να τονίσω. Πρώτον, εύρος και φύση των κυρώσεων. Δεύτερον, ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου <clears throat> και ως θεματοφύλακα των συνθήκων αλλά και αμερόληπτου πολιτικού οργάνου, ενός ένα αμερόληπτο πολιτικό όργανο θεσμικά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε.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 Thank you very much, President. πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Άκουσα και τους άλλους συναδέλφους και μένα με ανησυχεί το ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να μελετήσουμε το θέμα αυτό, σε αυτό το σχέδιο γράφω. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε γι' αυτό το λόγο να περιμένουμε πολύ για τα συμπεράσματα. Νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι συμφωνούν εδώ με τον κύριο στόχο που είναι να σώσουμε την Ευρώπη από την κρίση. Να βρούμε τρόπους και μέσα και το πλαίσιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μας επιτρέψουν να σώσουμε το ευρώ, να εγγυηθούμε ότι το ευρώ θα λειτουργεί σωστά και θα ξεπεράσει την κρίση. Νομίζω θα πρέπει να συμφωνήσουμε, θα πρέπει να αυξήσουμε τις ικανότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας της Ένωσης να καταστήσουν δυνατό κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα παρόλα αυτά να πω, με πολλούς άλλους συναδέλφους που είπαν ότι υπάρχουν ήδη πολλά μέσα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε περαιτέρω. Το Κοινοβούλιο προσφέρει στα πλαίσια των συζητήσεων πακέτου τέτοιου είδους μέσα. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσουν να βρούμε μια πρακτική λύση το όλο θέμα. Τώρα, στα πλαίσια Αλλαγή στις ε, συνθήκες με αυτέ αυτές τις αλλαγές νομίζω ότι μα απομακρύνει το στόχο μα να σώσουμε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχο τον οποίο επέλεξαν οι Πρωθυπουργοί και αργοί κρατών των κυβερνήσεων αλλά από νομική πλευρά, την άποψή μου είναι αμφίβολο ο τρόπο. Ε, με τον οποίο θέλουμε να χειριστούμε το πρόβλημα και δεν νομίζω ότι σε αυτή την ε, κατάσταση, σε αυτό το στάδιο θα μπορούσαν να ευρεθούν με αυτόν τον τρόπο απαντήσει τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, για τη συνθήκη. Βρέθηκε ένας τρόπος να προχωρήσουμε, αλλά δεν είναι ικανοποιητικός. Αρχίζοντας με το εξής. Πρώτα απ' όλα, το κάποια θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν στο περιθώριο, όπως το δικό μας. Ιδιαιτέρως. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας υποσχολεί πάρα πολύ όλους μας. Δηλαδή βασικά ο τρόπος με τον οποίο έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα αφήνει κατά μέρο τη δική μας, το δικό μας θεσμικό όργανο. Και αρχίζοντας, κάνοντας ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ξέρω πόσο μακριά μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υπάρξει προβλήματα και κρίσεις που έχουν σωθεί δημιουργώντα κάποια προηγούμενα. Αλλά τώρα, εάν αυτή η διακυβερνητική συνθήκη παίρνει ένα μεγάλο μέρος κυριαρχίας κάποιων κρατών μελών σε σχέση με την ε, αρχική συνθήκη που πάμε. Διότι η αρχική μας συνθήκη έχει τους τρόπους της, τις διατάξεις της. Λέμβανε πάντα υπόψη τις περισσότερες παραδόσεις και τις εθνικές νομοθεσίες με ειδικέ ε, διαδικασίες στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας και κράτος για να αλλάξει η συνθήκη. Όπως φερειπίνει το δημοψήφισμα. Και επιτρέψτε μου σε αυτή τη στιγμή να πω το εξή. Εδώ και κάποιους μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέκρινε το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας της, της συνθήκης. Και αν τώρα, μετά από τρεις-τέσσερις μήνες κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα χωρίς να κάνουμε τις κατάλληλες συζητήσεις, εμείς θα πρέπει να το επισημάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαφορετικά θα παίζουμε στην παγίδα των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ακόμη και αυτό το σύνταγμα, το οποίο επικρίθηκε τόσο πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εισαγάγει για πρώτη φορά μεταξύ των κρατών μελών το θέμα των συνταγματικών κυρώσεων τα οποία, και πολλοί μας έχουν πει τον τρόπο με τον οποίο βάλλονται οι κυρώσεις. Τώρα φτάνουμε στις κυρώσεις, θέμα το οποίο ανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι. Πώς θα συντονίσουμε τέτοιου είδους κυρώσεις στα πλαίσια της κάθε εθνικής ομοθεσίας, αν η πρώτη χώρα η οποία το έκανε στην δική, το δικό της σύνομα και που εισήγαγε αυτό το μέτρο το οποίο το έκανε για πρώτη φορά στη δική του ε, στη δικό του εθνικό δίκαιο και στη δική του νομοθεσία επικρίθηκε πριν από λίγες μήνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα βλέπουμε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς όταν κάνουμε τέτοιου είδους κρίσεις και κυρίως για αυτό το θέμα των κυρώσεων. Τώρα επανέρχομαι στο θέμα μας. Δεν είναι. Δεν έχουμε συνηθίσει με τέτοιου είδου, τέτοιου είδους προβλήματα να αντιμετωπίζουμε σε εθνικό επίπεδο. Και η χώρα με επικρίθηκε διότι είπε ο Πρωθυπουργό μα ότι θα ήθελε το θέμα αυτό να το ε, αναφέρει στο εθνικό του κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Το εθνικό κοινοβούλιο του καθενός, του οποίου έχει πιο περιορισμένες αρμοδιότητες και συνήθως από ό,τι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και σύντομα. Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω την ελπίδα ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπο με τον οποίο συνταγματικές λύσεις θα ευρεθούν και ξέρουμε ότι εμείς στην Επιτροπή μας να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και συμφωνώ με αυτό το οποίο ελέγχθη για την Οικονομική Επιτροπή. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το τυπικό, αν θέλετε, και εκείνοι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο. Πώς μπορούν οι στόχοι που θα τεθούν και θα θεσπιστούν από να υλοποιηθούν. Πιστεύω ότι πραγματικά με ψυχραιμία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα και την εργασία των επιτροπιακών. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Το συζητήσαμε. Το θέμα αυτό περίπου για μία ώρα και 20 λεπτά. Πρόκειται για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά έχουμε κάποιες ιδέες, ο καθένας εξέφρασε την απόψή του. Κάποιοι συνάδελφοι είναι υπέρ. Θα πρέπει να το σκεφτούμε το όλο το θέμα πολύ σοβαρά και κυρίως κατά τη διάρκεια των ε, διακοπών των Χριστουγέννων θα συναντήσουμε τους συναδέλφους αργότερα και θα μπορέσουμε συζητώντας μαζί τους να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθούμε. Θα ήθελα τώρα να περάσω στο επόμενο θέμα, η ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση του προηγούμενου θέματος θα συνεχιστεί στην κοινή συνεδρία. Το επόμενο θέμα αφορά εμένα. Είμαι εισηγητής. Τροποποίηση των άρθρων 87 και 88 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, η θέση ισχύ της συνθήκης Λισαξέ εκ βαθέων αυτό το οποίο καλούσαμε στο παρελθόν επιτροπολογία. Σήμερα η συνθήκη της Λισαβόνα, το άρθρο 280 και 90 ε, και 91 προβλέπει ότι θα μπορούν να νομοθετούν διανάθεσης κάποιων αρμοδιοτήτων οι χώρες, αλλά μιλούμε για νομοθετική πράξη και δίνουμε στην Επιτροπή την δυνατότητα να εκτελέσει μια πράξη η οποία της έχει ανατεθεί στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας. Βεβαίως, όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν εκ των υστέρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μπορεί να επιφέρει κάποιες αλλαγές και ή να ανακαλέσει αυτή την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης προς την Επιτροπή. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές στον κατανοησμό μας. Διότι το άρθρο 291 της Λισαβόνας προβλέπει την δυνατότητα για την Επιτροπή να εγκρίνει κάποιες εκτελεστικές ε, ε, πράξεις γενικού χαρακτήρα. Γενικού χαρακτήρα επαναλαμβάνω χωρίς να περιμένει να μεταφέρουν ε, στο εθνικό τους δίκαιο αυτές οι εκτελεστικές αρμοδιότητες επιτροπή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθά να ενεργούμε σε ορισμένε περιπτώσεις με ταχύτητα είναι αρκετά ε, απλό. Το σύστημα εγώ είμαι ο δικός σας εισηγητής, προτείνω να αλλάξουν τα άρθρα 87α ε, και 88, να έχουμε νέα ε, διατύπωση των άρθρων αυτών που θα αφορά τις πράξεις που αναθέτουμε και την διαδικασία κατά την οποία έχει θεσπίσει το Κοινοβούλιο μία βασική εκτελεστική ε, πράξη βάσει των σχετικών ε, διατάξεων του κανονισμού και συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 51. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται ότι όταν παραλάβει ο πρόεδρος κατά τη πράξη και εκτελεσής πράξης ε, την ε, νομοθετική πράξη, την διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή, ζητά να συντάξει η αρμόδια επιτροπή μια έκθεση και να δει κατά πόσον αυτή η διαδικασία είναι σωστή ή θέλει ακόμη και να την ανακαλέσει σε περίπτωση διαφωνίας. Αυτό γίνεται για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις. Και εδώ προβλέπεται η διαδικασία που έχουμε εμείς για τον έλεγχο, για την με ορισμό προθεσμίας εξέταξης, για έγκριση ή απόρριψη. Ή με μία επίσημη πράξη μπορεί να αποφασίσει ότι συμφωνεί και δεν έχει καμία αντίρρηση. Θα πρέπει να δούμε τώρα πώς στο σύνολό του θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε στο Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του για την όλη υπόθεση και την όλη πράξη που του δείτε να εξετάσει. Εάν ακολουθεί η συνήθι διαδικασία και φτάσει από την αρμόδια επιτροπή η έκθεση στην Ολομέλεια, κανένα πρόβλημα. Αν η τη ουσία αρμόδια επιτροπή δεν λάβει απόφαση στα πλαίσια της προθεσμίας που έχει οριστεί, ο πρόεδρος μπορεί να επαναφέρει το θέμα στη μερίσια διάρκεια Ολομελίας αν το ζητήσουν 40 ε, βουλευτές, υπάρχουν υπογραφές από κάποιες πολιτικές ομάδες. Έτσι, τελική απόφαση, ο διτητής αν θέλετε τελικά για την όλη διαχείριση του όλου θέματος είναι η Ολομέλεια. Και επίσης σε περίπτωση που αποφασίσει για μία κατατουξιοδότηση πράξη και αρμόδια επιτροπή εταίων εντάξει μπορεί ο πρόεδρος να αποφασίσει σύμφωνα με μία ταχεία διαδικασία, ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί. Το ίδιο ισχύει και με τις εκτελεκτιστικές πράξεις. Εδώ προβλέπεται ένα μεταβατικό καθεστώς, διότι η άσκηση των δικαιωμάτων ουσίας εκ μέρους της Επιτροπής υπόκεινα στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Ιουνίου 1989. Οι νομοθετικές πράξεις που θα υιοθετηθούν πριν από την θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού υπόκεινται σε αυτή την απόφαση και, σε και στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται ο προηγούμενος κανονισμός. Άρθρο 13 του κανονισμού 182-211, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάποια άρθρα προηγούμενου κανονισμού. Τώρα, σε περιπτώσεις στις οποίες το άρθρο 50 ή 51 του κανονισμού προβλέπεται οι διάφορες επιτροπές συνεργάζονται βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού και ο πρόεδρος αποφασίζει αν οι εκτελεστικές πράξεις και οι εξουσιοδοτημένες εκτελεστικές πράξεις θα ακολουθήσουν την διαδικασία που είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη θεώρηση του κανονισμού. Δηλαδή θα αποφασίζει ο πρόεδρος εάν τελικά στα πλαίσια του άρθρου 50 και βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται το όλο θέμα αυτό ανάλογα με τη φύση του θα ανατεθεί σε μία μόνο αρμόδια επιτροπή ή αν θα κληθούν περισσότερε επιτροπέ να συντονιστούν και να συνεργαστούν μεταξύ του. Στο caso è previsto che ci sia un accordo tra i presidenti, che ci sia una fissazione di eh, riunione della commissione congiunta. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε και πώ θα γίνει η συνεργασία μεταξύ των δύο προέδρων των αρμόδιων επιτροπών. Διαφορετικά δεν μπορέσει να υπάρξει μεταξύ τη συμφωνία. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αποφασίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με το άρθρο 50. όπου οι δύο επιτροπές εργάζονται χωριστά για την ε, εξέταση των ε, κατεξεκολούθηση πράξεων και των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων όταν πρόκειται για δύο διαφορετικό θέματα. Αυτά είναι τα δύο νέα άρθρα. Αυτό σας προτείνω, αυτές τις αλλαγές. Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να θέσουμε κάποιους κανόνες ώστε να μπορούμε να ε, διατηρήσουμε τον έλεγχο, να κάνουμε τον έλεγχο με ταχύτητα και να αναθέτουμε τον έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή για νομοθετικά θέματα, αλλά να μπορεί να παρέμβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σύνθεση ολομελίας αν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά ήθελα να πω και περιμένω να κάνετε τώρα εσείς τη σχολεία. Ε, ο κύριος Ντάφε, Πρόεδρε, έχετε δίκιο πρέπει να πω ότι για το πρόβλημα των εντεταλμένων πράξεων και εκτελεστικών πράξεων και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό το θέμα το Κοινοβούλιο προκάλεσε και προκαλεί προβλήματα για το σώμα. Πιστεύω ότι οι δικές σας προτάσεις αυτό που κάνουν είναι και αποσαφηνίζουν ταυτόχρονα αλλά και απλουστεύουν τις διαδικασίες, τις διεργασίες αυτές. Όμως πρέπει να το συζητήσουμε, να το συζητήσω και με τους συντονιστές της ομάδας μου, ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη πλήρης αντίδραση, ιδιαίτερα από τους συντονιστές ε, όσον αφορά τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές που επομίζονται το νομοθετικό, την νομοθετική κυριότερη ευθύνη και έχουν και μεγαλύτερη πείρα όσον αφορά αυτά τα προβλήματα από ότι εγώ. Ε, Σε ευχαριστούμε. Και φυσικά αναφέρθηκα με συνθετικό τρόπο ε, εν περιλήψη στη δική μου περιγραφή για αυτά τα θέματα. Δεν θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Τις τροπολογίες σας, στις τροπολογίες μπορείτε να υποβάλλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο κύριος Γκερέρο, ευχαριστώ πρόεδρε. Στο τελευταίο τμήμα αυτής της παρέμβασης ε, κάποιες ανησυχίες ε, δημιουργήθηκαν. Γιατί αν είναι εν περιλήψη συνθετική αυτή η παρουσίαση, όπως την χαρακτηρίσατε, δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει όταν, τι θα γίνει όταν θα ακολουθήσει το γραπτό, ε, το γραπτό κείμενο. Και σε σχέση και με την ε, Ιταλική σχολή και όταν έχουμε τέτοιο βάθος, ιδιαίτερα όταν έχουμε και αρμοδιότητα από πλευράς κριτού ή δικαστή αυτών των θεμάτων. Και σε σχέση με τις άλλες χώρες, όπως π.χ. στην περίπτωση της Ισπανίας, έχουμε τις κατεντολήν πράξεις τους νόμους κατεντολήν Δίνεται για παράδειγμα η εντολή να αναπτυχθεί κάποια δράση από πλευράς της κυβέρνησης. Και έτσι έχουμε την εντολή για αυτή την δράση και πέρα από αυτό το πλαίσιο και τον έλεγχο. Και τέλος, το Κοινοβούλιο εξετάζει αν αυτή η εντολή χρησιμοποιήθηκε σωστά υπό τους όρους που είχε θεσπίσει και καθορίσει το ίδιο το Κοινοβούλιο από πλευράς του. Εδώ έχουμε ένα διαφορετικό μας πρόβλημα σε σχέση με τις ε, κατεντολήν πράξεις. Ε, το Κοινοβούλιο διατηρεί μια συγκεκριμένη θέση μπορεί να ακυρωθεί, να ακυρωθεί η εντολή όπως ε, και αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Κασίνη είναι ο καθορισμός των διαδικασιών ώστε ακριβώς να μπορεί να υπάρξει έλεγχος στην εκτέλεση αυτής της εντολής, στις κατεντολήν πράξεις Εν πάση περιπτώσει στην εκτέλεση αυτών των πράξεων, στις ε, ε πράξεις ε, κατεφαρμογή, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι πολύ πιο αφηρημένος και γενικόλογος. Είναι πολύ λιγότερο σαφής σε σχέση με τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται, που είναι πιο ευαίσθητου χαρακτήρα, ας το πω έτσι. Και σε κάποιο βαθμό εξαρτώνται από το ότι η Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να υπομισθεί να ενστερνιστεί το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των κατεντολήν πράξεων ή αυτών των κατεφαρμογήν πράξεων εξ ονόματος ε, σκιώδους εισηγητού της ομάδας μου που δεν μπορεί να παραστεί απόψε, Βιτάλ Μορέιρα, επισημαίνει ότι γενικά συμφωνεί με τις προτάσεις ε, όπως έχουν διατυπωθεί από τον πρόεδρο Κασίνη από πλευρά του. Όμω θα επιθυμούσε ο ίδιο να απλουστευτεί κάτι, να απλουστευτούν κάποιε από τι διαδικασίε που καθορίζονται και προαναγγέλει ο ίδιο ότι θα καταθέσει τροπολογίε προ αυτό το στόχο για αυτή την απλούστευση. Ευχαριστώ. Βλέπω να υπάρχουν άλλε παρεμβάσει από μέλη. Θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας ότι πράγματι, πράγματι οι κάποιες δυσκολίες που αντιμετώπισα προέρχονται από το γεγονός ότι στο Ιταλικό δίκαιο το οποίο γνώριζα ήδη η ορολογία είναι διαφορετική. Και νομίζω και το ίδιο ισχύει και σε άλλα δίκαια, σε άλλες χώρες, ε, σε σχέση με, ε, για παράδειγμα, δικαιοδοσίες όσον αφορά εδώ το Κοινοβούλιο. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί επίσης να ανήκει και στο εκτελεστικό αυτή η αρμοδιότητα, αυτή η δικαιοδοσία, στο εκτελεστικό σκέλος <clears throat> σε σχέση με τον καθορισμό των διατάξεων από πλευράς ε, Κοινοβουλίου ή έχουμε και άλλες ε, δυνατότητες ή δράσεις ε, από πλευράς μιας κυβέρνησης σε σχέση με τη δραστηριοποίησή της με τέτοιου είδους κατεντολήν ή κατεφαρμογή πράξης και μπορούν να αρχίσουν να ισχύουν με κάποιε εξαιρέσει μέσα σε μια προθεσμία κάποιων μηνών. Όμως η συνθήκη τη Λισαβόνα χρησιμοποιεί διαφορετική διαδικασία. Λέει ότι οι κατεντολήν πράξεις δεν είναι νομοθετικές πράξεις. Και έχουμε τον αντίστοιχο, το αντίστοιχο άρθρο που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υιοθετεί, να εγκρίνει μη νομοθετικά μέτρα. Είναι θέμα του πώς καθορίζονται και πώς καθορίζονται αυτές οι μη νομοθετικές πράξεις που είναι γενικότερου χαρακτήρα ή πιο γενικό, σε ένα γενικότερο ευρύτερο πλαίσιο. Κάτι διαφορετικό από τις ε, κατεφαρμογή ε, κατεκτέλεση πράξης Εν πάση περιπτώσει το πιο σημαντικό από όλα αυτά ποιο είναι. Είναι αυτό το οποίο έχουμε εδώ ενώπιόν μας. Το άρθρο 290 λέει ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει αυτό το άρθρο ότι νομοθετικές πράξεις ρητά προβλέπουν και θέτουν όρους και προϋποθέσεις κατ' εντολήν πράξεων. Δηλαδή για το ότι μπορεί να αποφασίσει είτε το Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο για την εφαρμογή τους, για την μετάθεση αυτών των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν ε, με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε, αν δηλαδή για παράδειγμα δεν υπάρχουν ενστάσεις από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου ή Συμβουλίου και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά νομοθετικό έργο μπορεί να μεταθέτει κάποιες δικαιοδοσίες ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη. Πάντα υπάρχει μια καταληκτική ε, προθεσμία μέσα στην οποία το Κοινοβούλιο μπορεί στο εκτελεστικό σκέλος να μεταθέσει τέτοιου είδους αρμοδιότητες ή να εκφράσει ενστάσεις και αντιρρήσεις ως προς αυτό. Και ως όσον αφορά το Κοινοβούλιο, θα πρέπει οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να εμπλέκονται και να εποπτεύουν και να παρακολουθούν τα θέματα. Εδώ ακριβώς έγκυται η περιπλοκή, ο πιο σύνθετος χαρακτήρας. Η δεύτερη πτυχή είναι το ότι η κατεντολήν πράξεις που θα αφορούν την ίδια την ε, αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, αν εγκρίνει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, τότε προχωρεί αυτή η πρωτοβουλία. Διαφορετικά, αν υπάρχει ένσταση, πρέπει να δούμε ποια αντιμετώπιση, ποιας αντιμετώπιση θα τύχει η ένσταση. Τότε θα πρέπει η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ίσω να αποφασίζει ποια συνέχεια θα δίνεται. Ελπίζουμε όμως ότι αυτό δεν θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία ώστε να οδηγηθούμε σε μια, ε, το πω έτσι, μεγαλύτερη ε, χρονική διάρκεια ρύθμισης αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, δεν είναι νομοθετικό, νομοθετικό έργο η κατεντολήν πράξη. Είναι, ας το πω έτσι, κανόνες εκτελεστική η δράση όσον αφορά το εκτελεστικό. Τώρα η ορολογία όσον αφορά αυτές τις κατεντολήν πράξεις και το καθεστώς έχει όπως σας περιέγραψα όμως υπάρχουν πολλές περιπλοκές ε, είναι σύνθετος ο χαρακτήρας και για ένα μεταβατικό διάστημα ως για μια μεταβατική περίοδο η προσαρμογή αυτών των διεργασιών για τις κατεντολή ε, κατεκτέλεση πράξης ε, και και κατ' εντολή πράξης πρέπει να δούμε αν εφαρμόζεται το άρθρο 51 σε αυτές τις καταστάσεις ή όχι. Αυτή είναι η περιπλοκή κατάσταση στην οποία προσπάθησα να ανακεφαλαιώσω και έχουμε και κείμενο επ' αυτών. Θα έλεγα να θέσουμε προθεσμία καταληκτική αστροπολογία στην 26 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Αυτή θα είναι η προθεσμία. Και θα το εξετάσουμε το θέμα στι 28 Φεβρουαρίου. Συμφωνείτε? με αυτή την πρόταση. Δεν βλέπω να υπάρχουν ενστάσεις. Λοιπόν αυτό θα κάνουμε, αυτή τη συνέχεια θα δώσουμε. Το άρθρο 6 τώρα, στη συνέχεια, είναι ένα διαφορετικό θέμα, όμως και πάλι από πλευράς μου είμαι εισηγητής επ' αυτού, είναι η εκλογή αντιπροέδρων όσον αφορά, είναι κάπως ευθύ, απλό το θέμα. Ζητήθηκε από εμά να συντάξουμε γνωμοδότηση για μια τροποποίηση του κανονισμού. Στην περίπτωση που αν ένας ή περισσότεροι αντιπρόεδροι θα έπρεπε να αντικατασταθούν, να μπορέσουμε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει. Εμείς τον διορισμό ενός αντιπροέδρου αν μπορούμε με ε, εκλογή διαβοής να ρυθμίσουμε το θέμα ή αν υπάρχει ένας αντιπρόεδρος που πρέπει να αντικατασταθεί, να δούμε πώς θα μπορεί να γίνει. Και είπαμε εντάξει, ωραία, δεν θα πρέπει να δεν θα υπάρχουν προβλήματα γιατί για όλη την εκλογή όλων των αντιπροέδρων είναι δυνατόν να εκλέγονται διαβοής και ο πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει αν υπάρχει ένας και μόνο υποψήφιος για παράδειγμα αν αυτό θα πρέπει να ισχύει Και τότε με βάση αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαμε να προβούμε στην αντικατάσταση. Α, όμως είχαμε και το θέμα της, ε, του ότι έπρεπε να εξεταστεί το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος και να γνωμοδοτήσουμε, να συντάξουμε γνωμοδότηση, ίσως αν χρειαστεί και να προτείνουμε και τροποποίηση του κανονισμού, αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν αντιπρόεδρο που πρέπει να αντικατασταθούν. Εκεί περιπλέκονται κάπως περισσότερο τα πράγματα, επειδή ε, όπως έχουμε και το θέμα των ε, της εκλογής, οι υφιστάμενοι κανονισμοί, οι ενισχύοι κανονισμοί προβλέπουν ότι όλοι για όλα αυτά τα αξιώματα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη σειρά στην ε, εκλογή για την εκλογή αρκετών. Πρέπει να έχουμε αρκετούς υποψήφιους για να καλυφθούν τα κενά. Τέσσερις θέσεις που πρέπει να πληρωθούν τέσσερι υποψήφοι. Εντάξει, πρώτο ερώτημα, μπορούμε να ρυθμίσουμε διαβοή στην εκλογή τους. Ο κανονισμό λέει ναι, οι διατάξεις ε, ε, ε, επιτρέπουν την εκλογή διαβοή. Τι θα γίνει όμως με την σειρά όσον αφορά την εκλογή τους. Ήθιστε μέσω του αποτελέσματος της ψηφοφορίας να καθορίζεται η σειρά τους όσον αφορά το το αξίωμά τους. Μπορούμε να προβούμε σε διαβοής εκλογή, όμως θα έπρεπε να γίνει εκλογή στη συνέχεια με ψήφους, με την έκφραση των, της βούλησης των μελών ψηφίζοντας, για να γνωρίζουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκλογής του καθενός. Για να γνωρίζουμε ποιος έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων. Τώρα, Ποιο είναι το νόημα να γίνεται διαβοής ε, ε, ε, εκλογή όταν ούτως ή άλλως πρέπει να ακολουθήσει η ψηφοφορία. Μια και όμως έχουμε τη δυνατότητα της διεξαγωγής εκλογής, πρέπει να έχουμε μια διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα να καθορίζει τη σειρά αυτών των αντιπροέδρων αξιωματικά. Και τι τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει, τι γίνεται, πώς θα, θα ρυθμίζεται το θέμα αν σε μια ψηφοφορία για εκλογή αντιπροέδρων αν είναι ορθό να επιτρέψουμε με μία ψηφοφορία να ε, ρυθμίζεται το θέμα. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε πρόβλημα, διότι όσον αφορά την έκφραση ε, των μελών υπέρ κάποιου αντιπροέδρου ήταν ένα ποσοστό 5 ή 6% κατά μέσον όρο δεν θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός ψηφοφοριών προς ψήφιση των ε, υποψηφίων, διότι δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Ο κύριος Βίλαν ζήτησε όμως πρώτος τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Βίλαν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε για αυτή την εισαγωγή που κάνατε και για την, ε, το έγγραφο εργασίας. Καταρχήν για το σημείο 2 μπορώ να αναφερθώ σε αυτό. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα το οποίο τίθεται στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μέσω του κανονισμού. Όταν έχουμε τόσους υποψηφίους όσα αξιώματα πρέπει να πληρωθούν, αυτό αφορά τους αντιπροέδρους και τους κοσμήτορες, τότε μπορεί, μπορεί, δεν είναι τελεσίδικο, μπορεί διαβοής να εκλεγούν. Δηλαδή διαβοής συνενετικά εκφράζεται η συνένεση διαβοής του σώματος και είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου αν θα διαξαχθεί ψηφοφορία, γύρω ψηφοφορίας ή όχι. Είναι πολιτικού χαρακτήρα θέμα, πολιτική επιλογή. Δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να πει κανεί όταν μία αναγκαία, ένα αναγκαίο αριθμό, είτε μια κοινοβουλευτική ομάδα, είτε δύο, είτε 40 μέλη, πρέπει να γίνει μυστική ψηφοφορία. Η μόνη δυνατότητα θα ήταν αν μία ομάδα έλεγε τότε θα έχουμε και εμείς υποψήφιο από πλευράς μας Τότε λοιπόν θα είχαμε δεύτερο υποψήφιο και αυτό είναι πάλι κάτι ενδιαφέρον να βλέπαμε αυτή την προοπτική. Η πρόταση δική σας όμως πρόεδρε είναι θελκτική, μας θέλει επειδή ε, δεν δημιουργεί πρόβλημα θα πρέπει να υπάρχει κάποια απαρτία, κάποιος συγκεκριμένος αριθμός ή όχι. Θα πρέπει να γίνεται η ψηφοφορία και μπορεί να ακολουθήσει ψηφοφορία, η ουσιαστική έγκριση δίνεται διαβοής. Και αν χρειαστεί προβαίνουμε μετά σε μυστική ψηφοφορία και έχει το πλήρες δικαίωμα η Ολομέλεια να, κάνει, να προβεί σε αυτή τη ρύθμιση. Νομίζω πολύ επαρκώς αναφερθήκατε στο θέμα αυτό της εναλλακτικής αυτής δυνατότητας που θα δίνεται στην Ολομέλεια. Για το 2Β όμως το θέμα είναι πιο περίπλοκο. Και ειλικρινά πρέπει να πω δεν υπάρχει μία απάντηση που να ικανοποιεί απόλυτα. Το 2Β δεν αφορά μόνο την εκλογή αντιπροέδρων, αφορά και τους κοσμήτορες. Αφορά όλες τις εκλογές, εκλογικές διαδικασίες, όπου περισσότεροι υποψήφοι είναι υποψήφοι για την εκλογή ενός αξιώματος. Και έχουμε την αρχή πρώτος γύρος απόλυτη πλειοψηφία, δεύτερος γύρος απόλυτη πλειοψηφία μόνο στον τρίτο γύρο ψηφοφορίας η απλή πλειοψηφία ε, ε, ε, ισχύει ως αρχή. Και αυτό για να ρυθμίσουμε το θέμα των περισσότερων υποψηφίων ουσιαστικά θα έπρεπε τους ε, επικεφαλείς ε, υποψηφίους με ευρεία πλειοψηφία να τους εκλέγουμε. Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται τότε με απλή πλειοψηφία. Η πραγματικότητα τι δείχνει. Στον πρώτο και δεύτερο γύρο κάποιοι εκλέγονται. Στον τρίτο γύρο πρόκειται για μια τελική αντιπαράθεση. Και σε μια τελική αντιπαράθεση μόνο ε, ο στόχος είναι φυσικά η απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά δεν έχουμε κανένα κανονισμό που να διασφαλίζει ότι κάποιοι βουλευτές, οι βουλευτές θα πρέπει ένα συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών να εκλέγουν και έτσι έχουμε δύο διατάξεις του κανονισμού που αντιβαίνουν η μία ή στρέφεται η μία κατά της άλλης. Και αυτό που έχετε στο έγγραφο εργασία σας ότι οι ευρωβουλευτές εκλέγουν έναν και μόνο αυτό είναι μια ακραία περίπτωση. Η διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, έχουν, έχει, έχει περιγράψει τον κανόνα κατά κανόνα των εκλογών. Και έχουμε εδώ την περίπτωση δηλαδή του λιγότερου, του μικρότερου από 50%, δεύτερο, στο δεύτερο γύρο 4,6%. Ο μέσος ευρωβουλευτής δηλαδή πώς συμπεριφέρεται. Κανένα στους δύο πρώτους γύρους ψηφοφορίας δεν εκλέγεται και όλα μετατίθενται προς απόφαση, προς ρύθμιση στον τρίτο εκλογικό γύρο. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να πει στον πρώτο γύρο τρεις να εκλέγονται, στο δεύτερο δεν εκλέγεται κανείς και μετά όλα τα νομικά θέματα ρυθμίζονται, πρέπει να ρυθμιστούν μέσω της τρίτης εκλογικής αναμέτρησης. Και θα πρέπει να δούμε ότι και για τους αντιπροέδρους και τους κοσμήτωρες αν αυτό θα πρέπει να ισχύει. Κοίταξα και άκουσα οι δύο μεγαλύτερες ομάδες του σώματος έχουν εσωτερικές διατάξεις ότι το ίμιση των ψήφων πρέπει να χρησιμοποιείται εκάστοτε οι δύο μικρότερες ομάδες, δηλαδή μια ομάδα που έχει οι ποσοστώσεις σε σχέση με την, τις εκλογικές διαδικασίες, η άλλη ομάδα έχει το single transfer vote, Ιρλανδική προσέγγιση δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει. Κάθε υποψήφιος έχει έναν αριθμό που λαμβάνει και ε, για όλους τους υποψηφίους ε, λαμβάνεται αυτό προς ρύθμιση. Αυτό που πρέπει να αποφασίσει το κοινοβούλιο δηλαδή είναι, ας το πω έτσι, το πιο ε, απόμακρο από την κανονική του διαδικασία. Και εδώ θα πρέπει να δούμε στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση, αυτό δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν θα υπάρξουν μεταβολές. Όμως μακρό πρόθεσμα, όσο περισσότερο θα έχουμε πάνω από 15 υποψηφίους ή 14 υποψηφίους και θα πρέπει η σειρά με μυστική ψηφοφορία να καθορίζεται, τότε επαρκούν οι ίδιοι μηχανισμοί ή όχι. Έχουμε το ερώτημα, μήπως θα πρέπει να ανατρέξουμε στην λύση που έχουν και οι ομάδες, δηλαδή να, πρέπει να αναλώνεται ένα συγκεκριμένος αριθμός ψήφων στην ψήφιση αυτών των ε, υποψηφίων και εγώ θα έτεινα να υιοθετήσουμε την λύση των δύο μεγαλύτερων ομάδων. Δηλαδή κατά ελάχιστο το ίμιση των ψήφων να μπορούν να αναλώνονται στον γύρο αυτό. Θα το χαιρέτιζα να, να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν έχουμε πίεση χρόνου. Θα, ε, δεν μπορούμε ούτως ή άλλως να ε, το λύσουμε αυτό μέχρι τον ε, Ιανουάριο. Θα έχουμε την ευκαιρία ίσως να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα πέρα από τις ε, πληροφορίες σας από την ε, διοίκηση, από τους υπαλλήλους, να δούμε ποιο κριτήριο πρέπει να ισχύει σε σχέση με τις ε, διεργασίες εκλογής όσον αφορά τα σημεία τα οποία εσείς έχετε ως αφετηρία. Ευχαριστώ. Ναι, λέει ο πρόεδρος. Εγώ παρουσίασα ένα έγγραφο εργασίας για να έχουμε μια γενική συζήτηση. Πρέπει όμως να λάβουμε αυτή την προκαταρκτική απόφαση. Πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός, ναι ή όχι. Αν πιστεύουμε ότι όντως πρέπει, θα ορίσουμε άλλη ημερομηνία και τότε θα έχω υποβάλει λεπτομερή έκθεση. Αν αποφασίσουμε ότι δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί ο κανονισμός, θα αφήσουμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή. Ο συνάδελφος αναφέρεται ε, στο γεγονός ότι κατά την άποψή του πιστεύει ότι όντως πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ο κύριος Νταφ, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, συμφωνώ. Θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες αναφορικά με αυτό το θέμα. Τίθεται καταρχάς ε, το ε, θέμα της ε, διαβοής έγκρισης του υποψηφίου. Νομίζω ναι. ότι είναι ένας αναχρονιστικός, αν θέλετε, τρόπος ναι. εκλογής. Το σύνηθες θα ήταν να έχουμε μυστική ψηφοφορία. Αυτό θα ήταν το φυσιολογικό έτσι ώστε ε, κάθε αποκλίνουσα άποψη να μπορεί ε, να εκφραστεί. Και οι εποχές βεβαίως και ε, οποιαδήποτε άλλη ψήφος. Όλα αυτά αρμόζουν στην συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται σε ένα δημοκρατικό νομοθετικό σώμα. Θα έλεγα ότι εάν ένας πρόεδρος εμένα προσωπικά μου ζητούσε να εγκρίνω διαβοής ε, τον ορισμό οποιοδήποτε υποψηφίου θα με έφερνε σε κάπως δύσκολη θέση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που σήμερα πλέον έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δεν τίθεται κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσε κάλλιστα η μυστική ψηφοφορία να γίνει ο μοναδικός τρόπος εκλογής. και έτσι θα λύνονταν και όλα τα άλλα προβλήματα περί προηγουμένων και άλλα. Τώρα, ως προς τη μεθοδολογία, δική μου προτίμηση και προτίμηση της πολιτικής μου ομάδας είναι να αλλάξει το σύστημα το παρόν της ισόρευσης ψηφοφοριών και να μεταβούμε σε ένα ενιαίο ε, σύστημα, μία ε, ψηφοφορία πολύ πιο απλή, πολύ πιο δίκαιη, πολύ πιο ξεκάθαρη. Θα ήθελα να μου δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να επανέλθω σε αυτό το θέμα και να το αναλύσω ε, περισσότερο σε βάθος. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης ε, για το έγγραφο εργασίας και τις προτάσεις. Με τη σειρά θα τα πάρω. Στο πρώτο σημείο θα ήθελα να τοποθετηθώ που μετά γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όταν έχουμε τα άλλα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και καταλήγουμε σε μια τροποποίηση του κανονισμού αν χρειαστεί. Εγώ θεωρώ ότι η διαβοής εκλογή είναι μια έσχατη λύση, αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας. Το κοινοβούλιο, καλό είναι να μην εκλέγει διαβοής. Ήδη αναφέρθηκε από τον συνάδελφο. Εν τω μεταξύ μια ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν κρατάει τόσο πολύ, ούτε καν τόσο όσο μια άλλη. Όμως δημοκρατικά είναι, νομιμοποιεί περισσότερο μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Με πρότειναν μια φορά για ένα αξίωμα που διαβοής θα, εξε, θα εκλεγόμουν και είπα όχι, αρνούμε να το κάνω. Αυτή η ιδιαίτερη ευθύνη που θα είχα αν εκλεγόμουν σε αυτό το αξίωμα πρέπει να έχω τη βεβαιότητα ότι η πλειοψηφία των μελών θέλουν να με διορίσουν σε αυτό το αξίωμα με πλειοψηφία. Και έτσι έχουμε αυτό τον κανόνα ε, ε, ε, υπάρχει η, η ευτυχής ρύθμιση ότι έτσι ρυθμίζονται τέτοιου είδους θέματα και θα ήθελα με αυτόν τον τρόπο να ρυθμίζονται τα αξιώματα. Όταν προτείνονται κάποιοι υποψήφοι από τις κοινοβουλευτικέ ομάδες υπάρχει κύρος και βάρος σε αυτή την εκπροσώπηση για το κοινοβούλιο συνολικά και γι' αυτό θα πρότεινα συνολικά πάντα να εκλέγουμε να γίνεται η εκλογική διαδικασία και όχι να εκλέγουμε διαβοής. Τώρα, αν παραμείνουμε στην ερμηνεία που δόθηκε τον Ιούνιο, ότι παρεκκλίνοντας θα μπορούμε και διαβοής να εκλέγουμε σε κάποια αξιώματα. Τότε όμως κατεπηγόντως θα συνιστούσα, κατεπηγόντως το Κοινοβούλιο να έχει την δυνατότητα να παρεκκλίνει, να αποστασιοποιείται από αυτή τη διαδικασία όταν ε, δικαιολογείται, όταν για παράδειγμα 40 μέλη το απαιτούν ή μια κοινοβουλευτική ομάδα διαφωνεί. Θα ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση, μη ικανοποιητική και δημοκρατικά δεν θα μπορούσαμε προ τα έξω να δικαιολογήσουμε μια τέτοια κατάσταση στου πολίτε αν είμαστε ανήμποροι ω κοινοβούλιο και αναγκαζόμαστε να εκλέγουμε κάποιον ω αντιπρόεδρο που <coughs> δεν θα τύχαινε πλειοψηφία από το σώμα για να προτείνεται η εκλογή διαβοή. Γι' αυτό πιστεύω προσωπικά ότι όταν έχουμε τη διαβοή σε εκλογή, αν αυτό θα ήταν η επιθυμία και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει η ε, δυνατότητα έκφραση τη ένσταση, εν πάση περιπτώσει, εναντί μια τέτοια υποψηφιότητα μέσω μια ενισχυμένη μειοψηφία, λέγει ο μιλητή. Και για το σημείο 2α, μια καλή πρόταση που υποβάλλεται, διότι προτείνεται μια μυστική ψηφοφορία. Για το 2Β παρόμοια το βλέπω όπως και ο συνάδελφος Βίλαντ. Με τη μόνη διαφοροποίηση, τη μόνη διαφορά ότι για αυτή την εκλογική διαδικασία, όπως κατάλαβα και τον κύριο Μακντάφ, ότι την single transferable vote, την μία αλλά ε, με δυνατότητα μεταφοράς ε, ψήφο, στη ψηφοφορία θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. Δηλαδή σε σχέση με τον υποψήφιο που θα έπρεπε να αναδειχθεί αν δεν υπήρχε καλύτερη διαδικασία ανάδειξης, όμως υπάρχει μια καλύτερη διαδικασία ανάδειξης του αλληλότερου υποψηφίου και αυτής πρέπει να κάνουμε χρήση. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκερέρο παρακαλώ. Πρόεδρε, πολύ σύντομα ευχαριστώ για να επισημάνω ότι πιστεύω ναι ότι πρέπει να τροποποιήσουμε τον κανονισμό και πιστεύω επιπλέον ότι είναι καλό, είναι θετικό να μην είναι ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου που θα αποφασίσει τη σειρά όσον αφορά την τους αντιπροέδρους ε, γιατί δεν είναι μια προεδρικού χαρακτήρα ε, ένα, ένα προεδρικού χαρακτήρα θεσμικό όργανο και παρότι υποβάλλονται υποψηφιότητες από τις κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει να βασίζονται στην υποστήριξη των ευρωβουλευτών οι υποψήφοι και πρέπει να διαφοροποιείται η δυνατότητα έκφρασης αυτής της υποστήριξης ανάλογα με την κάθε υποψηφιότητα που εκλέγεται και το αποτέλεσμα ψήφων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να καθορίζεται από το αποτέλεσμα το εκλογικό η σειρά τους και όχι από απόφαση του Προέδρου. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε κύριε Γκερέρο. Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι που να έχουν ζητήσει τον λόγο. Και νομίζω λοιπόν ότι από αυτούς που σχολίασαν προηγούμενα φαίνεται ομόφωνα να ακολουθείτε η τάση, να εκφράζετε η τάση ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε τους ε, κανόνες. Ε, μια ριζοσπαστική προσέγγιση, παστική πρόταση να έχουμε μία ψηφοφορία που εντάξει μπορεί να μην είναι ομόφωνη ως προς αυτό το σκοπό αλλά ο κύριος Φίλαντ υπέβαλε μία πρόταση. Ένας ελάχιστος αριθμός πρέπει να καθορίζεται που θα πρέπει να ισχύει. Εν πάση περιπτώσει θα διατυπώσουμε, θα συντάξουμε μια πιο εξειδικευμένη ε, έκθεση στις οποίες ε, θα, στην οποία θα μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες <coughs> ώστε να μπορέσει να εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη προς έγκριση δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι τόσο περίπλοκο, δεν έχουμε την πίεση χρόνου εξάλλου κατά τα άλλα είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που θα έπρεπε να έχουμε επαρκή χρόνο για να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Νομίζω μπορούμε να επανέλθουμε το Φεβρουάριο με την έκθεση, αν συμφωνείτε. Και με αυτέ τι παρατηρήσει μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7. Ο συνάδελφο Ντάφ είναι εισηγητή. Είναι μια έκθεση που έχει υποβάλει με βάση το άρθρο 172 και ζητά ε, να καταστεί υποχρεωτική ονομαστική ψηφοφορία. Ε, στην τελική ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή ή στην Ολομέλεια. Θα πρέπει λοιπόν η τελική ψηφοφορία να είναι ονομαστική όταν πρόκειται για την τελική έγκριση. Έχετε το λόγο κύριε Ντάφ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι ε, ξεκάθαρη η πρότασή μου. Βελτιώνεται ξεκάθαρα η δημοκρατική πρακτική. Καθίσταται περισσότερο διαφανής και αναγνωρίζουμε το ότι ο νομοθετικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά με την συνθήκη της Λισαβόνας και αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχουν οι επιτροπές στη γενικότερη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που η διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης μας αφορά όλο και περισσότερο και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίσταται ουσιαστικός νομοθέτης και ειδικότερα βέβαια οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πιστεύω ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να υιοθετήσουμε αυτή την πρακτική εάν πραγματικά φιλοδοξούμε να φτάσουμε ε, σε όσο δυνατόν υψηλότερο επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας. Θα πρέπει λοιπόν να είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία όταν έχουμε να κάνουμε με νομοθετική διαδικασία στις επιτροπές. Και θα πρέπει τα αποτελέσματα να καταχωρίζονται στα πρακτικά, ακριβώς όπως ε, γίνεται και με την Ολομέλεια. Από εκεί και πέρα, σκέφτηκα επισταμένος ε, τι θα γίνει με την αλλαγή αυτή στη διαδικασία. Το σκέφτομαι το θέμα από τότε που υπέβαλε το πρώτο σχέδιο διατύπωσης. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συμπεριλάβουμε το άρθρο 166 και το άρθρο 167 στη δεύτερη του παράγραφο στο 196. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Στη συνέχεια θεώρησα ότι η πιο ξεκάθαρη ε, προσέγγιση θα ήταν για όλους μας να τροποποιήσουμε το άρθρο 195 και να προσθέσουμε εκεί ένα εδάφιο το οποίο να, να λέει το εξής. Όταν γίνεται ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής για μια συγκεκριμένη νομοθετική πράξη, όποια και να είναι ε, η φάση της διαδικασίας που ε, ε, σημειώνεται εκείνη τη στιγμή, κάθε τέτοιου είδους ψηφοφορία λοιπόν θα είναι ονομαστική. Και γι' αυτό το λόγο έχω υποβάλει τρόπο, μία τροποποίηση, μία πρόταση τροποποίησης της δικής μου Έκθεση. στη δική μου έκθεση μάλλον. Και αυτό το έκανα σήμερα το απόγευμα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Προς το παρόν, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγνιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άντριου, είναι σημαντικό να μπορώ να πω ότι μερικές φορές συμφωνώ μαζί σου. Το λέω για να γνωρίζουν όλοι ότι γίνεται και αυτό. Δυόμιση χρόνια βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βλέπουμε να γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες σε τροπολογίες όχι τόσο σημαντικές και τελικά δεν έχουμε ονομαστική ψηφοφορία στην έγκριση του τελικού κειμένου το οποίο ουσιαστικά είναι και το πιο σημαντικό νομοθέτημα. Θα πρέπει ε, τα μέλη των εκλογικών μας ε, περιφερειών ε, να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς ψηφίσαμε στην τελική ψηφοφορία του εκάστοτε κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Ανταλλάξαμε ρόλους με τον κύριο Άγνιου σήμερα. Βρίσκω πιστικά αυτά τα οποία ήθιστε να και παρουσιάζει ο κύριος Αντριού ε, Νταφ. Σήμερα όμως όχι. Δεν μπορώ να κατονίσω γιατί σε όλες τις φάσεις πρέπει να την πρόταση αυτή σε σχέση με τη διαβούλευση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή όλα ε, με ονομαστική κλίση, με ονομαστική ψηφοφορία να ρυθμίζονται. Ούτε για την Ολομέλεια δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Μπορεί να ζητηθεί, αλλά δεν είναι δεσμευτικό ως αρχή, εν πάση περιπτώσει. Βλέπω μια αξιοπερίεργη σύμπτωση λοιπόν αυτού του αιτήματο, αυτής της δυνατότητας με αυτό που σήμερα με την έκθεση του κυρίου Γκερέρο που έχουμε στο τραπέζι για συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης να προβλέπονται οι δυνατότητες το κοινοβούλιο λέει για άλλη μια φορά να ψηφίζει και για τροπολογίες και τέτοιες προτάσεις και άλλες προτάσεις που στοχεύουν τις διονομαστικής ψηφοφορίας ψηφοφορίες να τις περιορίσουν. Ενώ ο Άντρου Νταφ λέει κάθε ψηφοφορία για νομοθετική πρόταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει με νομαστική ψηφοφορία να ρυθμίζεται. Πρέπει σχετικά με, με, με, κάποιο πραγματισμό, με κάποιο ρεαλισμό να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν αυτές οι διαδικασίες για όλα τα στάδια της εξέτασης να ε, προβλέπονται. Και ενώ για την Ολομέλεια θα ήταν ε, μεγάλο ε, έλλειμμα αν την ανάγκη αυτού του χρήσιμου μέσου την δίναμε στα, ε, στις κοινοβουλευτικές ομάδες ε, και ε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαμε να αποκαταστήσουμε την, ε, ας το πω έτσι, το κύρος των εργασιών μας. Ακόμα δεν έχω πλήρως πιστεί. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, μια και ακούσαμε και τα υπέρ και τα κατά ως επιχειρήματα. Και είναι, δεν είναι κάτι ασήμαντο το θέμα αυτό, παρότι στην αρχή όταν άρχισα την εξέταση αυτού του θέματος φαινόταν ότι ήταν κάτι το εύκολο να ρυθμίσουμε. Όμως τα επιχειρήματα εξακολουθούν και υπάρχουν όπως και πριν. Και θα ήθελα λοιπόν να πω και εγώ αυτό το οποίο ανέφερε ο προλαλή ότι έχουμε κάποιο χρόνο που μπορούμε να τα, πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Η ομάδα μου θα ήθελε να συζητηθούν αυτά τα θέματα στο μέλλον τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και να επανέλθουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά τον κύριο Χέφνερ αναφέρθηκε στο σχέδιο έκθεσής μου για το άρθρο 70. Αυτό το οποίο ορίζεται εκεί είναι το εξής. Άπαξ και έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, η Επιτροπή υποχρεούται να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Δεν λέει όμως ότι είναι απαραίτητο η ψηφοφορία αυτή να είναι ονομαστική. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Νταφ, να πω ότι όντως είναι σημαντικό να συζητηθεί το θέμα αυτό στις ομάδες μας, στις πολιτικές, να πάρουμε το σφιγμό. Θα έλεγα ότι στη δική μου πολιτική ομάδα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος ε, ε, ό,τι έχει να κάνει με τη διαφάνεια αυτό το μητρό διαφάνειας, έτσι όπως το αποκαλούμε. Οι συνάδελφοί μου πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αμοιβαία απάντηση, ανταπόκριση από πλευράς Κοινοβουλίου, να είναι το Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο. Να φανεί ξεκάθαρα ότι όταν αποφασίζουμε ε, και νομοθετούμε ουσιαστικά, ε, είμαστε υπόλογοι πολιτικός και δημοσίως ε, αποδίδουμε το λογαριασμό. Κάνουμε αυτό το, αυτή την άσκηση λογοδοσίας. Εκπλήσωμαι διότι βλέπω ότι ενδεχομένως άλλες ομάδες δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή επιμένοντας την ονομαστική ψηφοφορία σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να το ζητήσουν το 1 τέταρτο των μελών. Αυτή είναι μια διαδικασία αρκετά άκαμπτη και καλό θα ήταν να ε, ρυθμιστεί. να εξυγχρονιστεί. Αυτό είναι ό,τι πιο εξυγχρονιστικό πιστεύω μπορεί να κάνει ένα σύγχρονο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Καλώς. Προχωρούμε λοιπόν. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι 26 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν συμφωνείτε κύριε Ντάφα. Ο κύριος Ντάφ. Νομίζω ότι επειδή είπαν συνάδελφοι ότι θέλουν να το συζητήσουν στις πολιτικές τους ομάδες, καλύτερα να ε, θέσετε την προθεσμία για το Φεβρουάριο, κύριε Πρόεδρε, ούτως ώστε να μπούμε στον κύκλο του Φεβρουαρίου σε επίπεδο ε, επιτροπών για να υπάρξει περισσότερος χρόνος. Κανένα πρόβλημα, λέει ο Πρόεδρος. Καλώς. Επομένως, ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών θα είναι 28 Φεβρουαρίου το μεσημέρι και άρα στην επόμενη συνεδρίαση μετά από αυτό ε, θα έχουμε την ψηφοφορία. Καλώς, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε φτάσει στις 6.30 που είναι η ώρα κατά την οποία ε, θα διακόψουμε, αλλά έχουμε ολοκληρώσει την ε, εξέταση της ημερήσιας διάταξης. Νομίζω ότι μπορούμε να διακόψουμε λοιπόν για μία ώρα περίπου, διότι στις 6.30 θα ξεκινήσουμε ε, με την κοινή συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση της δικής μας Επιτροπής 25 Ιανουαρίου του 12 από 3 μέχρι 6.30 και 26 Ιανουαρίου του 12 από τις 9 μέχρι τις 12.30. Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30. Εκεί θα πρέπει να αποφασίσουμε για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση αυτή, αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και ε, τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, ο υποφαινόμενος δηλαδή, ε, θα σας πει τι θα ε, κάνουμε άπαξ και λάβουμε τις απαντήσεις τους. Θα πρέπει να υπάρχει πιο συγκεκριμένη εντολή από τη διάσκεψη των Προέδρων. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε ορίσει ε, την ημέρα ε, αυτή, 9 Ιανουαρίου. Είναι ανοιχτή ακόμα η μερίσια διάταξη μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Διακόπτουμε μέχρι τις 6.30. Ευχαριστώ.